Let me see my Greek. I don't have my Greek. Anyway, I'll No, now it's here. Ε, καλή, καλή σας μέρα. Καλημέρα, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Χουντή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, δεν προτίθεμε. συζητάμε το θέμα της ε, επικαιροποίησης της γνωμοδότησης της επικαιροποίησης συγγνώμη, της οδηγίας που έχει τον τίτλο ε, αυτό δεν συζητάμε που έχει τον τίτλο της επιδράσεις των δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Είναι η τέταρτη φορά που κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Επομένως, κυρία Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω ό,τι έχω πει στις αρχικές τοποθετήσεις, ούτε αυτά που περιλαμβάνονται στο κείμενο το οποίο έχετε μπροστά σας και περιμένω τις τροπολογίες. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα θα πω δύο πράγματα ενημερωτικά για να δείξω τη σημαντικότητα του θέματος αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο είναι ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συζητώντας την υπόθεση του αεροδρομίου του Σάλτσμπρουκ κατέληξε ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις ενός σχεδίου στο περιβάλλον ώστε να αποφεύγεται η παράκαψη του στόχου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τη σαλαμοποίηση, δηλαδή κατά τεμάχη ας πούμε των σχεδίων, αλλά να αξιολογούνται στο σύνολό τους. Είναι μια παρατήρηση που μας είναι μια απόφαση του δικαστηρίου που μας είναι πολύ χρήσιμη όσο αφορά την επεξεργασία της δικής μας πρότασης. Και το δεύτερο ενημερωτικό που θέλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι είναι το γεγονός ότι στο Συμβούλιο, πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος συζητήθηκε το θέμα και περισσότερο δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην απλοποίηση της διαδικασίας και όχι στη βελτίωση της ποιότητας. Εδώ... to be silent. Thank Λέω το δεύτερο είναι η πρόσφατη, απόφα... η πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος έδωσε, συζήτησε το θέμα, αυτό που μας αφορά, και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην απλοποίηση της διαδικασίας και όχι στη βελτίωση της ποιότητας. Εδώ έχουμε βέβαια μια αναγνώριση των κρατών μελών ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται σωστά, υπάρχουν ανεπάρκειες, αλλά αυτό το θέμα της διαδικασίας με περιθώρια περισσότερης ευελιξίας είναι που όπως έχουμε διαπιστώσει που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως, στο σημείο αυτό όπου τίθεται από την πρόταση της Κομισιόν, όπως έχουμε πει και σε άλλες ε, συζητήσεις μας, οι δικές μου προτάσεις είναι να το περιορίσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται ευελιξία, εξαιρέσεις που δημιουργεί, ε, όπως δείχνει η εμπειρία, πολλές, ε, πολλά προβλήματα. Οι άλλες παρατηρήσεις μου έχουν να κάνουν ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εφαρμογή της οδηγίας και λόγω ενδεχομένως της κακής εφαρμογής και ούτω καθεξής και η συμμετοχή του κοινού ε, ήταν ε, ανύπαρκτη έως ανεκτή. Ε, αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα κράτη έχουν κινηθεί με διαφορετικό τρόπο. Επομένως η οδηγία και η δική μας η πρόταση πρέπει να ομογενοποιήσει την εφαρμογή της και να είναι πιο αυστηρή όσο αφορά αυτά τα, θέματα. Δεν θέλω να σας κουράσω καθόλου παραπάνω. Θεωρώ ότι το κείμενο αυτό που θα διατυπώσουμε εμείς και βεβαίως η έκθεση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να προλαμβάνει και όλα αυτά για τα οποία έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές και για άλλη μια φορά σημειώνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Τα επίκαιρα στοιχεία που σας έδωσα είναι για να δείξουν και τη σημαντικότητα του θέματος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κουντή. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος να κάνει κάποια παρέμβαση, Περιμένουμε. Α, παρακαλώ την Επιτροπή. Ναι. Ο κύριος Κλέμνης. Ο κύριος Κλέμνης. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Χουντή ε, και για τις παρατηρήσεις του και για το μέχρι σήμερα έργο του. Επιτρέψτε μου να περάσω στην ε, lingua franca. I wanted on behalf... Θα ήθελα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Χουντή και να πω το εξή, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το σωτερευτικό αποτέλεσμα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην πρότασή μας στο παράρτημα 3. Εκεί αναφερόμαστε στη σώρευση και με άλλα έργα αλλά και με άλλες δραστηριότητες, projects και activities. Είπαμε ε, αναφερόμαστε και στα δύο αυτά. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Τώρα όσον αφορά την δημόσια την συμμετοχή του κοινού ε, Βεβαίως χαιρετίζουμε κάποιες βελτιώσεις που έκανε ο κύριος Χουντής ε, στην πρότασή μας και που θα ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι το Συμβούλιο μέχρι τώρα δεν άνοιξε τη συζήτηση για διατάξεις που δεν καλύπτονται από την πρόταση της Κομισιόν και θα L δεν θα θέλαμε να διευρύνουμε τη συζήτηση σε άλλα θέματα όπως προτείνει ο, ο κύριος Χουντή σε άλλα θέματα δηλαδή που δεν καλύπτονται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχουν καθόλου συζητηθεί με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ο, περιορίστηκε σε αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Φοβάμαι ότι αν διευρύνουμε τη συζήτηση θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Και βεβαίως ε, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Δεν, θα, εκείνο που θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν είναι να μην χρησιμοποιηθεί σαν πρόσχημα η πρόταση αυτή για να ανοίξει συζήτηση άρθρων που δεν έχουν, που δεν καλύπτονται από την πρόταση της Επιτροπής. Αυτό θα πάρει πολύ χρόνο επίσης και αυτό δεν το θέλουμε. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις. Περιμένουμε την έκθεση του κυρίου Χοντή και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε αν θέλετε την νομοθετική διαδικασία αν θέλουμε να ε, έχουμε αποτελέσματα. Αυτών λεχθέντων υπάρχουν βεβαίως πολλές τροπολογίες που κατέθεσε ο κύριος από πλευρά του κυρίου Χοντή. Σε γενικές γραμμές τις βλέπουμε θετικά. Θα τις δούμε θετικά σε επόμενα στάδια. Κύριε Βοστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις. Καλώς ορίζω την πρόταση του αγαπητού συναδελφού, του κυρίου Κουντή. Και είμαι πολύ ικανοποιημένο καταρχήν με τις δικές του συνεισφορές και να προσθέσω και με τον αγώνα για μια ανεξάρτητη εταιρεία που θα προβεί στη μελέτη αντικτύπου. Και ξέρω ότι ακόμη και η Κομισιόν δεν ήταν τόσο ικανοποιημένη, ακόμη και το Συμβούλιο δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο. Θα πρέπει ακριβώς να καθορίσουμε τις ε, προϋποθέσεις υπό ε, τις οποίες θα λειτουργήσει εντελώς ανεξάρτητα αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Και εγώ θα ζητήσω περαιτέρω διευκρινήσεις από τον εισηγητή, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και ότι ποτέ δεν θα ε, μπορέσουν ούτε οι διοικητικές αρχές ούτε οι πολιτικοί να αμφισβητήσουν ε, τη δουλειά αυτών των εμπειρογνωμόνων. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος να κόψουμε τους δεσμούς μεταξύ του επενδυτή και της εταιρείας ε, που καλείται να προβεί στην περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Και κάτι ακόμη. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με την πρότασή του όταν περιορίζει και διευκρινίζει δύο πτυχές. Τα project που μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου, τα οποία πρέπει να μπουν με σαφήνεια σε ένα κατάλογο να αποσαφινιστούν, χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερο περιθώριο λιγμό στα κράτη-μέλη. Όμως εδώ θα πρέπει να ξαναπούμε ότι όταν αυτά τα έργα σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα, πρέπει να δούμε ότι η δημόσια συμμετοχή θα πρέπει να περιοριστεί για να μην μπορεί να απαγορευτεί τελείως. Επίσης, η συμπερίληψη της διασενοριακής ε, τυχής στην μελέτη αντικτύπου. Ήταν ο κρίκος που έλειπε μέχρι σήμερα και τώρα και με τη δική μας συνεισφορά και της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος θα είναι κάτι σχετικό για το μέλλον και την ε, δημοσία συμμετοχή. Πρέπει να είναι δεσμευτική, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ειλικρινά ε, θα γίνει αυτή η συμμετοχή, δεν θα καλέσουν κάποιοι τους φίλους τους αλλά όσοι πραγματικά φύγονται από το θέμα αυτό θα πρέπει να ακουστεί η φωνή τους και θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και στη συνέχεια δεν μπορούμε να καλέσουμε για περαιτέρω συνεδριάσεις γιατί τελικά θα γίνει σχεδόν αδύνατη διαδικασία. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει διαφάνεια στην όλη διαδικασία ότι όλες οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται και θα είναι προσβάσιμες με κάθε διαθέσιμο μέσο, αλλά να μην έχουμε συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων και συναντήσεις επί συναντήσεων, γιατί Δεν νομίζω ότι χρειάζεται οι συμμετέχοντες ή εμπλεκόμενοι στο project να συναντιούνται κάθε εβδομάδα και επίση θα ήθελα να καλέσω μια συνεδρίαση ε, με τους σκιώδεις εισηγητές προκειμένου να αποσαφινιστούν ε, κάποια σημεία και κατόπιν να αρχίσουμε να συνεισφέρουμε και με τροπολογία στην εξαιρετική αυτή έκθεση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και παρακαλώ σημειώστε ότι υποστηρίζουμε πλήρως την προσέγγισή σας ε, και την έκθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Uh, We uh, expect your final Περιμένουμε το τελικό σχέδιο κειμένου. Η προθεσμία είναι 7 Μαΐου. Παρακαλώ κύριε Χουντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο για τα σχόλια που έγιναν ε, από τους συναδέλφους, ο κύριος Μποστινάρου. Περιμένω, θα κάνουμε τη συνάντηση, περιμένω τις, περιτέρω, ε, τις τροπολογίες, ώστε να το αποσαφηνίσουμε τι θέλουμε και να το κάνουμε. Πρόθεσή μου και ελπίζω πρόθεση των συναδέλφων είναι η Επιτροπή μας να φτιάξει ένα ισχυρό κείμενο για να μπορεί να έχουμε ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα. Στον αγαπητό εκπρόσωπο και συμπατριώτη από την ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν στο θέμα που έθεσε για άλλη μια φορά ότι η έκθεσή μας, η δική μας γνωμοδότηση ανοίγει και άλλα θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνει η αρχική πρόταση της Κομισιόν και ενδεχομένως ή μάλλον και δεν περιλαμβάνεται και στα όσα συζητάει το Συμβούλιο θέλω να του πω βεβαίως το γνωρίζει πρώτον ότι το, το, το τι συζητάει ή τι θέτει ως θεματολογία η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταρχήν δεν δεσμεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο, ε, από όσο ξέρω και η Επιτροπή Περιβάλλοντος κινείται σε αυτή την ευρύτερη θεματολογία. Δηλαδή το ανοίγει το θέμα, ανοίγει και άλλα θέματα και νομίζω ότι πρέπει να τα ανοίξουν. Τώρα και τελευταίο, τώρα ε, το αν ανοίξουμε και άλλα θέματα <clears throat> παραπέμπει στο ότι θα ανοίξουμε το κουτί της πανδώρας ή ε, έχοντας μια τέτοια μπορώ να πω ότι στο τέλος το κουτί της πανδώρας είχε την ελπίδα. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν η Επιτροπή και το Συμβούλιο βεβαίω να ακούσει τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη δική μα Επιτροπή και να τα κάνει τα πράγματα όπω νομίζουμε, όπω θα ισχυριστούμε εμεί ότι είναι καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω ότι έχετε δίκιο στο θέμα αυτό. Μπορούμε να ανοίξουμε όσα θέματα θέλουμε. 7 of May, 7th of May for our amendments to the rapporteur. 7 Μαΐου είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες μας προς τον εισηγητή. Team concerning... Προχωρούμε. Uh, uh, possible errors and omissions in the... Προχωρούμε στο θέμα υπαριθμών 17 για το πιθανά λάθη για το γραμματικό. Που έρχομαι εδώ. Σας θυμόμαστε. Μας θυμάστε. <laughs> Και εγώ σας θυμάμαι. θα μιλήσουμε για το γραμματικό, για τη διαχείριση των απορριμμάτων. θα μιλήσω στα ελληνικά. Έχω φτιάξει ένα presentation, ένα PowerPoint, και θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στον κύριο Απαζή από την προηγούμενη συνεδρίαση ότι ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 1988 να συζητείται, έγινε νόμος του κράτους το 2003 και αυτόν πάνε να υλοποιήσουν αυτή τη στιγμή. Όμως τότε ήταν κυβέρνηση σοσιαλιστική, η κυβέρνηση του Πασόκ, ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ, σοσιαλιστική, με πολλά στελέχη όμως της τότε σοσιαλιστικής κυβέρνησης κατηγορούνται σήμερα για διαφθορά. Και αυτό πάμε να συζητήσουμε σήμερα. Ένα μικρό παράπονο, αν θέλετε, στην Επιτροπή αναφορών σχετικά με την απάντηση που έλαβα στις 30 Μαΐου όσον αφορά α, α, σημείο που λέει ότι α, αν, εν πάση περιπτώσει, μια ομάδα κατοίκων δεν είναι σύμφωνοι με το σχέδιο, όσο σκληρό και αν είναι, ε, αυτό πρέπει να γίνει γιατί έχουν, ε, γίνει, πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ληφθήσεις από τη δικαιοσύνη αποφάσεις. Η δικαιοσύνη παραπλανήθηκε όμως και για το γραμματικό και για πολλά άλλου χιτά. Π.χ. καρβουνάρι. Υπάρχουν ψευδή στοιχεία. Α, το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ΠΕΣΔΑ, Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, είναι οι υπερδιαστολογημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης σύμπτων απορριμμάτων, mixed, mixed waste. Μιλάμε για σύμπτα απορρίμματα, τύπου χιτά φυλής. Οι πανομοιότυπες προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ, Αττικής, για κερατεία και γραμματικό, είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα προφανούς ασυμπατότητας με την κείμενη νομοθεσία αλλά και με την κοινή λογική. Ανάλυση του κ. Δημήτρη Δαμάσκου, μηχανολόγου μηχανικού. Και σε όλα αυτά έχει να, έχει να προσθεθεί και ένα τελευταίο, η απόφαση σταθμό 20-2012 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Στην διαφάνεια αυτή θα δείτε τα αποτελέσματα α, το 2007 σε σχέση με, τις, με το σύνολο των 27 χωρών όσον αφορά στην ανακύκλωση. Η Γερμανία πρώτη, σε πρώτη θέση είναι η Γερμανία, τότε έρχεται η Γερμανία, η Ολλανδοί, οι Σουηδοί, οι Δανείοι. Ε, η ε, τέταρτη θέση από το τέλος, 24η θέση, έρχεται η Ελλάδα. Και χώρες όπως η Κύπρος, η Πολωνία, η Λιθουανία που γίνανε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, α, λογικό είναι να έχουν την τελευταία θέση. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε τα αποτελέσματα, αυτά, αυτά είναι τα αποτελέσματα του 2012, Όσο αφορά με την ανακύκλωση και τον τρόπο που επιλέγει κάθε χώρα να διαχειρίζει τα απορρίμματα. Τελευταία η Ελλάδα. Πρώτη έρχεται η Αυστρία, οι Ολλανδοί, οι Δανείοι. Τελευταία έρχεται η Ελλάδα και μας έχουν ξεπεράσει χώρες όπως η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που έγινε μέλος το 2007, η Ρουμανία, 2007 και οι υπόλοιπες χώρες. Αυτό δεν δημιουργεί ένα ερώτημα. Τι γίνεται επιτέλους στην Ελλάδα. Γιατί ε, τόσα χρήματα έχουν δοθεί, ε, τόσες επιδοτήσεις ε, όλα αυτά τα χρόνια για να γίνουν υποτίθεται έργα ανάπτυξης, για να γίνει ανακύκλωση. Γίνεται ανακύκλωση. Τι γίνεται. Η Κομισιόν τι απαντάει σε όλα αυτά. Και περιμένω προφανώς μια απάντηση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, και αυτό είναι και, είμαι, και χαίρομαι που είναι ο κύριο Κρεμλής εδώ και ίσω πάρω μια απάντηση γιατί έχω στείλει επιστολή στον κύριο Κρεμλή, δεν έλαβα ποτέ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κρεμλής στην εφημερίδα Καθημερινή στις 19 του 2012, μίλησε για αλλαγή μοντέλου στη διαχείριση των απορριμμάτων που εξετάζει η Κομισιόν. Ισχυρίζεται μεταξύ των άλλων ο Κρεμλής πάντα με τη συνέντευξη τύπου που έδωσε τότε, ότι το έργο αυτό των των απορριμμάτων όπως επιχειρείται να δημοπρατηθεί, χρειάζεται σχεδόν το 100% των απορριμμάτων που παράγονται στην Αττική. Άρα μηδέν ανακύκλωση. Μηδέν ανακύκλωση. Αυτό να τονιστεί, ώστε να δικαιολογήσει φαραωνικά έργα για τη διαχείρισή τους. Λίγους μήνες αργότερα, ο κύριος Κρεμλής, όπως και εκπρόσωποι από την Γενική Διεύθυνση, από την Γενική Διεύθυνση από την Task Force, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, βρίσκονται στην Ελλάδα συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου του 2012 και ε, συμφωνούν στην κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων απορριμμάτων στην Αττική. Μεταξύ αυτού ένα είναι και στο γραμματικό, στην Κερατέα και δύο στη Φιλή. Και ε, θα ήθελα να μάθω, ε, θα ήθελα να πάρω μια απάντηση από τον κύριο Κρεμλή, γιατί αυτή η αλλαγή στάσης, πού οφείλεται. Ε, και όλα αυτά την ώρα, είδαμε στις διαφάνειες προηγουμένως, η Πορτογαλία το 2007 ήταν στη 15η θέση, το 2012 ανέβηκε στη 15η θέση και όλα αυτά την ώρα που ακόμα η πρόσφατη έκθεση με αριθμό 20 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2012 θέτει σε αμφισβήτηση τη χρηματοδότηση υποδομών επεξεργασία σύνδεκτων απορριμμάτων. Σύμφωνα με τι υποδείξει του κ. Δημήτρη Δαμάσκου, μηχανολόγου μηχανικού, έχω στείλει τα στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και περιμένουμε απάντηση όσον αφορά για την Ελλάδα. Αυτή είναι η απάντηση που παραλαβείς από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Dear Mr. Gikas, I acknowledge receipt of your emails dated 260213 and 120413, including the annexes, and inform you that your correspondence is currently being assessed by the Competence Auditing Chamber. I will inform you of the outcome of their assessment as soon as possible θα uh, will be able to do, will be able to that with the next four weeks. Σε τέσσερις εβδομάδες ε, θα μάθουμε και την απάντηση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά για τη διαχείριση των ε, απορριμμάτων ε, στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση αναφορά δεν πρέπει να μείνει, πρέπει να μείνει ανοιχτή και πρέπει να περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα στην Κομισιόν είναι τι έχει κάνει μέχρι σήμερα για υποτίθεται τις οργανωμένες χωματερές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε να υποστηρίξω ότι ένας χαδάς, μια ανεξέλεγκτη χωματερή, δεν πρέπει να κλείσει. Οι χαδά πρέπει να κλείσουν. Και αυτοί μπορούν να κλείσουν μια ανοιχτή. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Μπορούν να κλείσουν με ανακύκλωση, με, μια, με ένα ε, σωστό management, με μια σωστή οργάνωση. Από εκεί και πέρα Πάμε να δούμε ε, πολύ λίγο, πολύ γρήγορα, τι έγιναν σε άλλες περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα στο χιτά Σάμου, στο, στο χιτά Φιλής, στο Καρβονάρι, στη Μαυροράχη και στο γραμματικό που πρόκειται να φτιαχτεί. και ε, ακόμα δεν λειτουργεί. Χιτά Φιλής, ο μεγαλύτερος σκουπιδότοπος της Ευρώπης. Η χαρά των δημάρχων και η χαρά των εργολάβων. Το τι χρήμα κατασπαταλήθηκε όλα αυτά τα χρόνια για το χιτά πιστεύω ότι δεν θα μας φτάσουν ε, συνεδρίες για μήνες να συζητάμε και πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο ε, χιτά. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δώσατε εσείς κύριοι χρήματα για το συγκεκριμένο χιτά να γίνει ένα εργοστάσιο παλιά βέβαια αυτό, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Το φτιάξατε σε μια περιοχή η οποία στην πλαγιά ενός βουνού και στη συνέχεια έγινε κατολιστήσεις και το εργοστάσιο αυτό καταπλακώθηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ, όμως ο Ευρωπαίος πολίτης πλήρωσε το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Γι' αυτό η Κομισιόν τι έκανε. Α, δεν υπήρχε πρόδειλο σφάλμα. Και επίσης θα ήθελα έναν από τους ε, εκπρόσωπους της Κομισιόν να μου δώσει τον ορισμό, τη σημασία του πρόδειλου σφάλματος. Γιατί κάπου, δεν, ε, κάπου αυτό μέχρι τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε την ερμηνεία. Ένα ακόμα, και το, αυτό το παραδείχθηκε ο κύριο Γουρό και ζήτη, απολογήθηκε γι' αυτό, για τους καρκίνους που έχουν αυξηθεί, για τις α, για τα καρδιακά. Ο κόσμος πεθαίνει εκεί. Χιτά φιλή, ο μεγαλύτερος σκουπιδότοπος της Ευρώπης και κανείς δεν μιλάει. Οργανωμένος χιτά με τις ευλογίε της Ευρωπαϊκή Ένωση. Χιτά μαυροράχη. Ε, η μόνηση τεράστια και ε, σε, ε, με αποτέλεσμα να μολύνεται η αποξηραμένη ε, λίμνη Κορώνια. Τι έκανε η Κομισιόν γι' αυτό, δεν δίνεται εκεί πρόδειλα ασφάλματα. Οι αθεόφοβοι πήγαν και φτιάξανε χιτά στη Σάμο επάνω σε σαθρό έδαφος. Με αποτέλεσμα, κατά τη λειτουργία του χιτά στη Σάμο, αυτό, τα απορρίμματα όταν γέμισε να μετακινηθούν, και να πάνε όλα στη θάλασσα. Η Κομισιόν τι έκανε για αυτό το χιτά στη Σάμο. γιατί οι μέχρι τώρα απαντήσει που λαμβάνουμε από την ε, Κομισιόν είναι ότι παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας συνίσταται μόνο στην περίπτωση που το σχέδιο αρχίσει να εκτελείται χωρίς να συμφο... συμμορφούνται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η εν λόγω νομοθεσία για το περιβάλλον. Τι κάνατε κύριοι της Κομισιόν για το χιτά Σάμου. Πήγαν και φτιάξαν χιτά στη θέση που λέγεται βυθίσματα. Και μόνο η τοποθεσία δεν τους έλεγε τίποτα. Χιτά Λευκίνης. Παρακαλώ, ε, ναι, καταλαβαίνω το, τη σημασία όσων λέτε, αλλά επειδή ο ναι. χρόνος δεν είναι απεριόριστος και επειδή μιλάμε για το γραμματικό... Για το γραμματικό. Πάμε στο γραμματικό. Έρχομαι στο γραμματικό. Γραμματικό. Πήγαν και φτιάξανε, χωροθέτησαν χιτά πάνω σε ρέματα. Α, αυτό ε, δεν είναι κάτι το οποίο ε, το λέμε εμείς οι κάτοικοι, η ομάδα των κατοίκων. Είναι αυτό που έρχεται βάσει με έγγραφα που απέκρυψαν. Οι εικόνες είναι από τις καταστροφές που γίνονται κάθε φορά που, ε, γίνονται, που, βρέχει. Η παραλία σε γραμματικού ε, γίνεται καφέ από τη λάσπη που ξεκινά από το χώρο του χιτά και κατευθύνεται και, και χύνεται μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι απαθείς κοιλάδες κύριε Κουνιώτη, είναι ρέματα και ε, εδώ είναι μια αλληλογραφία που έχω με τις δραστηριότητες αγροτικές που αναπτύσσονται στην περιοχή. Το προσπερνώ. Αυτό το έγγραφο είναι έγγραφο της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής το 2005 το οποίο δείχνει, φαίνεται ότι στην περιοχή εκεί υπήρχαν δύο ρέματα που εκκινούν από την περιοχή του Χιτά που έχει χωροθετηθεί και καταλήγουν στη θάλασσα. Μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε μελέτες με πανεπιστήμια, γνωστά όλα αυτά θα σταθώ στο πόρισμα των ε, επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ε, έγιναν καταγγελίε, Εγώ από την Αγγλία πρώτος έκανα την καταγγελία από τη, ε, στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Προ τιμή ο Γενικός Διευθυντής, ε, ο κύριος Παναγιώτης Μέρκος, ξεκίνησε τη διαδικασία με αυτοψία στο χώρο, πήγαν οι επιθεωρητέ περιβάλλοντος. Έχουμε το τελικό πόρισμα. 18 Πρώτου 2012 πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος που αποδεικνύουν τα ατοπήματα, τις παραλήψεις στην ε, εν λόγω περιοχή. Επαναλαμβάνω κύριε Κογινιώτη, δεν είναι απαθείς χιλάδες, είναι ρέματα, όπως είχατε απαντήσει την προηγούμενη φορά. Και παρακαλώ μια απάντηση σε αυτό το έγγραφο. από εκεί και πέρα, οι κάτοικοι προσπάθησαν να κάνουν γεωτρήσεις. Έχουμε προσπαθήσει δύο φορές να κάνουμε διερευνητικέ γεωτρήσεις και μας σταμάτησαν οι ελληνικές αρχές. Γιατί αυτό δεν είναι πρόδειλο σφάλμα. Τι κάνει η Κομισιόν για αυτό το θέμα, κύριε. Α, και θα σταθώ σε αυτό, προτού τελειώσω. Α, θα, θα το διαβάσω αργά για να μπορέσουν οι μεταφραστές να σας το μεταφράσουν. Έχουν, έχω επανειλημμένα ζητήσει να ενημερωθώ για τον φορέα ή την αρμόδια υπηρεσία που εξέτασε την πληρότητα της συγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Μεταξύ των απαντήσεων που έχω λάβει, ενδιαφέρον προκαλεί η απάντηση της ΕΙΠΕΙΠΕΚ, Υπουργείο Περιβάλλοντο, η οποία αναφέρει επιλέξει «Η αξιολόγηση γεωλογικών μελετών δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας». Ε, επαναβάλλω, η μόνη υπηρεσία που μπορεί να ελέξει είναι αυτή. Αλλά αυτοί απαντούν, η συγκεκριμένη υπηρεσία, ότι δεν είναι αρμοδιότητα τη υπηρεσία μα. επαναλαμβανω η μονη υπηρεσια που μπορει να ελεξει ειναι αυτη αλλα αυτοι απαντουν η συγκεκριμενη υπηρεσια οτι δεν ειναι αρμοδιοτητα τη υπηρεσία μα. Επίση, υπαρχει πλεον και επισημα η ομολογια τη ΕΙΕΠ, δημόσια αρχή, για την αδειοδότηση της ΟΕΔΑ σε κοινοβουλευτικό έλεγχο όπου κατέθεσαν ότι δεν ήταν και δεν είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της γεωλογικής υδρολογικής μελέτης η οποία ήταν επισυναπτώμενη στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή η ομολογία καταρρύπτει τόσο την επιστημονική όσο και την νομική εγκυρότητα της διαδικασίας χωροθέτησης του έργου που επικαλείστε. Ο λόγος είναι ότι η ομολογία αυτή αποκαλύπτει ότι το πέμπτο τμήμα του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την έκδοση των αποφάσεων 1952 2007 και 1951 2007, που ουσιαστικά επικαλείστε, οχυρώνεστε κύριοι της Κομισιόν πίσω από αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραπλανήθηκε από την αδειοδοτούσα αρχή, διότι βασίστηκε στην απόφαση στην απόφασή του σε τυπικό μόνο έλεγχο θεωρώντας η ουσία έχει εξεταστεί εντελεχώς από το ΙΠΚ. Και η απάντηση που έχω λάβει από την ίδια, από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι ότι ε, κύριε Γκίκα δεν ε, είμαστε υπεύθυνοι για το ε, έλεγχο ε, των διερευνητικών γεωτρήσεων. Εδώ δεν υπάρχει κύριε πρόδειλο σφάλμα. Με, η αναφορά που έγινε στις προηγούμενες αναφορές έγινε για το τι γινόταν στο παρελθόν. Και εδώ έχουμε ένα οικολογικό έγκλημα όπως έγινε και στο παρελθόν. Δεν παραδειγματιστήκατε δεν υπάρχουν υποψίες από πλευρά της Κομισιόν. Θα οχυρωθείτε βέβαια από την απόφαση 85337 που λέει ότι κύριε εμείς δεν μπορούμε να ε, παρέμβουμε, ε, οι ε, γερμανικές εταιρείες δεν μπορούν να ελέγξουν τις ελληνικές, οι ελληνικές τις ιταλικές και ούτω καθεξής. Υπάρχει σε περιπτώσει μια γραφειοκρατία με τα αποτελέσματα και η οικολογική καταστροφή τεράστια. Α, από εκεί και πέρα, και τελειώνω με αυτό, η χώρα μου βρίσκεται σε ένα μνημόνιο κακός ή κακό δεν θα το συζητήσουμε σήμερα, και έχουν γίνει και πρόκειται να γίνουν μεταρρυθμίσει για να πληρωθεί ένα χρέο. Το νοικοκύρεμα και οι σωστέ μεταρρυθμίσει πρέπει να ξεκινήσουν από τη διαχείριση των απορριμμάτων για να εξοικονομηθούν χρήματα. Υπάρχει κόσμο που αυτοκτονεί λόγω του μνημονίου. Χάνονται περιουσίε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν ένα νοικοκύρεμα στα απορρίμματα. υπάρχει σταθμό 20, 20 του 2012 απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου από εκεί και πέρα, στην ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του γραμματικού υπάρχουν πρόδειλα σφάλματα, σοβαρά σφάλματα. Το έργο πρέπει να σταματήσει. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Κίκα. Νομίζω ότι είναι άμεση ανάγκη να συνεχίσουμε με την Επιτροπή. Ο κύριος Κουνινιώτης. Ναι. ναι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι ύψης της σημασίας και πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις που να εξασφαλίζουν μια ορθή διαχείριση, προκειμένου όχι μόνο να προστατευτεί το περιβάλλον, αλλά και η δημόσια υγεία. Η παρούσα αναφορά είχε συζητηθεί το Δεκέμβριο του 2011 στην Επιτροπή σας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τότε, αλλά και μέσω της συμπληρωματική απάντησης που απέστειλε το Μάρτιο του 2012, απαριθμίσει τους λόγους για τους οποίους δεν τίθεται θέμα παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα των οδηγίων 9931 <clears throat> περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 2008-98 για τα απόβλητα και 2011-92 ε, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων. Η Επιτροπή είχε εξάλλου, όπως είχαμε ενημερώσει, ανοίξει το 2004 και το 2008 δύο φακέλους προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση στο γραμματικό και είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχει ζήτημα παραβίαση. Η Επιτροπή <clears throat> δεν έχει λάβει καμία νεότερη πληροφορία που να μπορεί να αποδείξει μια δεχόμενη παραβίαση και να αντικρούσει τους <clears throat> ισχυρισμούς της. Ω εκ τούτου δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο θέμα αυτό, αλλά να σα ενημερώσω για την πορεία των διαφόρων υποθέσεων ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Όπω σα είχαμε ενημερώσει το Μάρτιο του 2012 για το θέμα του χιτά γραμματικού, του χώρου υγειονομική ταφή απορριμμάτων δηλαδή, έχουν ήδη εκδοθεί τρει αποφάσεις δικαστικές. Δύο από το Συμβούλιο τη Επικρατεία το 2007 και το 2012 και μία από το Γενικό Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όλες ήταν υπέρ της συνέχισης του έργου. Εκκρεμούσε επίσης μια υπόθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ωστόσο, στις 10 Ιουλίου 2012, το εν λόγω Πρωτοδικείο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κατατεθεί από κατοίκους και φορείς του Δήμου Μαραθώνα και αφορούσαν την κατασκευή του ΧΙΤΑ και το δικαστήριο έδωσε έτσι τη δυνατότητα να συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής. Ο Δήμος Μαραθώνα και διάφοροι φορείς της περιοχής κατέθεσαν αμέσως νέες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μία αίτηση αναστολής και μία αίτηση ακύρωσης του έργου. Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ωστόσο το αίτημα του Δήμου που ζητούσε την έκδοση προσωρινής διαταγής για πάγωμα της, προ... της προκήρυξης του διαγωνισμού, προκήρυξη που αφορούσε τη μελέτη, την κατασκευή και, και τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Η συζήτηση της κυρίας προσφυγής, δηλαδή της αίτησης ακύρωσης του έργου, είναι να πραγμα... ή μάλλον ήταν να πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2003. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμη αν έχει αναβληθεί αυτή η δίκη ή όχι ή... και δεν ξέρει πότε αναμένεται μια τελική απόφαση από το ΣΤΕ. Ωστόσο πρέπει να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι το ίδιο το Συμβούλιο έχει ήδη απορρίψει παρόμοιες αιτήσει το 2007 και το 2012. Οπότε αν όπως λέει ο αναφέρον είχε παραπλανηθεί το, το ΣΤΕ σε αυτές τις υποθέσεις, μάλλον τώρα θα λάβει μια σωστή απόφαση. Ε, σε αυτό το στάδιο θα ήθελα επίση να, επισημάνω δύο θέματα. Ε, πρώτον, ε, δεν γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η χωρητικότητα και η δυνατότητα του χιτά που είναι να κατασκευαστεί στο γραμματικό. Ο ανταγωνιστικό διάλογο είναι να γίνει αυτή τη στιγμή θα κατατεθούν οι προσφορές και τότε μόνο θα ξέρει κανείς γιατί μέγεθος μιλάμε. Γιατί βέβαια τα απορρίμματα δεν θα είναι ό,τι παράγεται θα μπαίνει στο χιτά, θα γίνει και μια ανακύκλωση και μια ανάκτηση. Ε, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα βέβαια, ε, δεν θέλω να επεκταθώ, βέβαια σε αυτό γιατί μίλησα για διάφορους ε, χιτά ανά της επικράτειας. Ε, θα ήθελα απλώς να πω η Επιτροπή τι κάνει, μας, μας ρωτήσανε. Πρώτον, ο σχεδιασμός δεν είναι θέμα της Επιτροπής είναι των ελληνικών αρχών να αποφασίσουν πώ θα σχεδιάσουν για να έχουν τι εγκαταστάσει τι εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια. Εδώ έχουν, ο Πεσδά αναφέρεται σε τέσσερι ε, χιτά. Αυτό είναι σεβαστό. Ε, ναι, από τέσσερι συγγνώμη. Ε, βέβαια, κανεί δεν απαγορεύει στην ελληνική δημοκρατία αν θέλει να αλλάξει το, σχεδιασμό και αντί για χιτά στο γραμματικό να κάνει εργαστήριο καύση με ανάκτηση. Αυτό δεν είναι θέμα τη επιτροπή. Πρώτο θέμα. Τι κάνει η Επιτροπή όταν λαμβάνει μια καταγγελία για δυσλειτουργία ενό χιτά, ερευνάει αμέσως και έχουμε πρόσφατα και πολλές υποθέσεις του καρβουναδίου που έχουμε ανοίξει φάκελο παραβίαση. έχουμε και διάφορες, δεν θέλω να επεκταθώ. Ε, θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο και για αυτή την υπόθεση, ότι στι 21 Φεβρουαρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταθέσει νέα προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της ελληνικής δημοκρατίας βέβαια, για το θέμα των, της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεκτης <clears throat> διάθεσης απορριμμάτων, δηλαδή των ΧΑΔΑ, και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών προστήμων. Στη περίπτωση που το δικαστήριο δικαιώσει την Επιτροπή, η ελληνική δημοκρατία θα οφείλει όχι μόνο να καταβάλει ένα συνολικό πρόστιμο για την παραβίαση, αλλά και επίσης ένα ποσό ημέρα μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης με την οποία ε, κάθε μέρα δηλαδή που θα συνεχίσει την παραβίαση. Και προκειμένου να σταματήσει αυτή η παραβίαση δεν πρέπει απλά να κλείσουν οι, οι χωματερές, η χαρά δηλαδή, αλλά τα απόβλητα που πήγαιναν μέχρι τότε στους χαρά να πάνε σε εγκαταστάσεις νόμιμες. Μία από αυτές είναι και το γραμματικό. Θα ήθελα, ε, τελειώνοντας, δύο απλά πολύ σύντομα, ε, Είχαμε επίσης και ένα έγγραφο ε, του, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στοιχεία 453.194 ε, και εδώ όπως το έγγραφο είναι στα αγγλικά θα αλλάξω γλώσσα, οπότε για τους μεταφραστές well, the, the document of 15 of September 2011 entitled Waste Management in Europe. Το έγγραφο αυτό που αναφέρεται στη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη και στις βέλτιστες ε, πρακτικές είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Γενική Νοματεία Ιστορικών Υποθέσεων και λέει διαθέσιμες ναι. πληροφορίες προτείνουν ναι. ότι η ε, οχήτα δραματικού είναι σημαντικές ε, προσπάθειες για να διορθώσουν την κατάσταση που προκαλείται από την κακή διαχείριση αποβλήτων. Φαίνεται ότι οι αρχές προσπαθούν να βρουν και να εφαρμόσουν εφαρμόσουν την καλύτερη λύση για ένα δύσκολο πρόβλημα με έναν τρόπο που να συνάδει πλήρω με την τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι θα κλείσω τα ελληνικά. Τελευταίο σημείο ε, έχουν αναφερθεί σε διάφορε συζητήσει η ύπαρξη διαφόρων μελετών που καταλήγουν σε διάφορα συμπεράσματα. Ε, βέβαια έχουμε εδώ δύο αποφάσει του Συμβούλου τη Επικρατεία που τι έχει αναλύσει όλε αυτέ. Εγώ μπορώ επίση να δώσω και μια άλλη μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το οποίο καταλήγει ότι, λέγοντας ότι όχι μόνο το, το, γραμματικό, το έργο του γραμματικού είναι κατάλληλο, αλλά αντίθετα υποστηρίζει μάλιστα ότι, ότι ο μεγάλος κίνδυνος υφίσταται από την κατέρευση του έργου, το οποίο παραμένει ημιτελές και δεν λειτουργεί. Σας ευχαριστώ. Εγώ κύριε Κουνιώτη, ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, προηγείται ο κύριος Χουντής. Ναι. Έχω το λόγο ή... Έχω το λόγο κυρία Πρόεδρε ή κάποιος συνάδελφος είπε επιπροσωπή. Έχω το λόγο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται να κυριαρχεί κυρια προεδρε η γλώσσα σήμερα, αλλά χθε είχαμε τα ισπανικά, έτσι λοιπόν. Πολύ. Θα αναφερθώ στην υπόθεση, θα είμαι, θα είμαι σύντομος παρακολουθώντας τη συζήτηση πια. Δηλαδή τους ισχυρισμούς που προέβαλε ο πρόσωπος τη ε, της Κομισιόν. Ε, η βάση, το, έργο το έχω δει και το έχω δει και σε κρίσιμες στιγμές, δηλαδή την ώρα της νεροποντής και επιβεβαιώνω την εικόνα που μας έδειξε από τις διαφάνειες ο κύριος ε, Γκίκας. Ε, αυτή είναι η εικόνα που εμφανίζεται μετά. Αλλά αυτό είναι ο λόγος, δηλαδή το έργο του γραμματικού και η προβληματικότητά του, που θα επισκεφτεί η Επιτροπή μας στην Ελλάδα. Η Επιτροπή και με τις σημερινές απαντήσεις αρνείται να τοποθετηθεί επί της ουσίας στο κεντρικό θέμα τουλάχιστον που θέτει η αναφορά του κυρίου Παπαδηγενόπουλου που αναφέρεται εδώ 573-2011 αρνείται δηλαδή να παρεύει που στο σημείο όπου διαπιστώνονται πρόδειλα σφάλματα. Αυτό το ξεπερνάει. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος αν θέλετε που μπορεί να παρεύει. Όχι αν λειτουργήσει το έργο και μετά από τη δυσλειτουργία θα παρεύει η Επιτροπή είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε στην έκθεση και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με συνέπεια να μην απαντάει σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα, τα έθεσε και ο κύριος Γκίκας, τα θέτει και η αναφορά, τα λέω και εγώ γρήγορα. Πρώτον, υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας όταν επεκτάθηκε η ισχύ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρχήν έγινε το 2003 και η επέκταση έγινε το 2009. Εμείς ισχυριζόμαστε και τεκμηριωμένα ότι δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία της κοινοτικής νομοθεσίας στην επέκταση αυτής της άδειας. Δεύτερον, και εδώ είναι το πολύ κρίσιμο και το επανέλαβε ο, εκπρόσωπος της Επιτροπής, εδώ δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε μόνο με μια τυπική γραφειοκρατία. Επικαλέστηκε αποφάσεις δικαστηρίων. Μα το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όλες αυτές οι αποφάσεις των δικαστηρίων, το λένε οι ίδιες, δεν έχουν μπει στην ουσία της υπόθεσης. Δεν έχουν μπει στην ουσία της υπόθεσης. Εξετάζουν τη διαδικασία της υπόθεσης. Επομένως, η τέτοια τοποθέτηση, να μου επιτρέψετε να σας πω, ότι είναι παραπλάνηση της Επιτροπής δεν υπάρχουν αποφάσει επί της ουσίας της υπόθεση στο δικαστήριο. Επομένω η επίκληση τη διαδικασία είναι παραπλανητικό. Δεν ε, λύνει το πρόβλημα όσον αφορά την... Ε, θα τελειώσω. Τρίτη παρατήρηση, υπάρχει έκθεση του, των επιθεωρητών περιβάλλοντο Μέσα στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται τη επίσκεψη να δούμε και αυτού του ανθρώπου που επιβεβαιώνουν αυτού του συγχειρισμούς. Και το τελευταίο είναι, ε, το θέμα είναι αφού διαπιστώνουν ή η Επιτροπή αφού υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα γιατί δεν απαντάει συγκεκριμένα και δεύτερο τι κάνει προκειμένου να αποτρέψει τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν στο έργο. Το επιχείρημα ότι οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για τη χωροθέτηση δεν αφήνει, δεν ξεπερνάει το πρόβλημα ότι η Επιτροπή έχει, έχει, είναι ευθύνη της εφόσον υπάρχουν πρόδειλα σφάλματα, εφόσον υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, να παρέμβει. Διαφορετικά, ξαναλέω, έχουμε να κάνουμε τουλάχιστον με μια δυσκίνητη γραφειοκρατική αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Δεν θα τα αναφέρω γιατί είναι πολλά. Στην περίπτωση της Ελλάδας τα ανέφερε ο κύριος Γκίτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Αν προτείνετε βέβαια την κατάργηση του έργου, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε στην Ελλάδα, όχι εδώ. Κύριε Χουντή, παρακαλώ, ο ναι, ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, the, ε, Οι αρμοδιότητες στη Γενική Διάθεση Περιβάλλοντος είναι του κυρίου Κουρνιώτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνω το λόγο για να απαντήσω σε κάποια πράγματα που είπε ο κύριος Γκίκας. Όπως γνωρίζετε το πρόβλημα με τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα που ε, ανάγεται στην εποχή προ μιας δεκαετίας. Ε, ο νόμος μετά το νόμο του 2002 και του 2006 ορίζονται ορισμένα πράγματα αλλά τελικά η, ο πληθυσμός ή οι τοπικές κοινότητες δεν δέχονται την α, ε, κατάσταση των τις τέσσερις εγκαταστάσεις που προβλέπονται σε εκείνο τον νόμο. Δεν δέχεται να γίνουν οι εγκαταστάσεις αυτές. Εμείς δεν ξέρουμε εάν μπορούμε να παρέμβουμε. Υπάρχουν επιχειρήματα του στυλ, η Δυτική Αττική λέει δεν μπορούμε εμεί να διαχειριζόμαστε τα πόλη τη Ανατολική Αττική η οποία δεν κάνει τίποτα. Εν περιπτώσει, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα ε, έργο. Τέσσερις προκηρύξει διαγωνισμών έγιναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα οριστούν ποσότητες εγώ αυτό που είπα για το 100% δεν σημαίνει ότι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης. Θα φροντίσουμε να είναι αυτό το πρώτο που θα εγκριθεί. Και ο στόχος για την ανακύκλωση μέχρι το 2020 είναι 50% και αυτό πρέπει, είναι νομική υποχρέωση αυτή ε, η οποία πρέπει να τηρείται για αλουμίνιο, γυαλί, ε, πλαστικά κτλ. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αγνοήσουμε την ανακύκλωση. Από οι στόχοι της ανακύκλωσης πρέπει να τηρηθούν. Προς το παρόν όμως, δεν, προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει ε, φόβος ότι οποιαδήποτε εργοστάσιο, οποιαδήποτε κατάσταση δεν θα ανταποκριθεί στους στόχους και από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν ακόμη συζητήσεις για τα ποσά, για τις ποσότητες αποβλήτων. We Επίσης, Ε, το θέμα της ανακύκλωσης είναι κάτι στο οποίο επιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια. Έχω πει στον κύριο Γκίκα ότι είναι, προσπαθούμε να δώσουμε τις διαφορετικές σακούλες στα διάφορα νοικοκυριά για να γίνεται η ανακύκλωση. Όμως δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να κάνουμε την ανακύκλωση και δεν μπορούμε να επιμένουμε στην ανακύκλωση άμα τα σκουπίδια είναι στο δρόμο και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μεγάλη εγκατάσταση καύσης στη φυλή στα λιώσια να καίμε τα σκουπίδια για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια αυτό γίνεται σε άλλες χώρες όπως παραδείγματος χάνει στο Βέλγιο ενδεχόμενα αυτό να είναι μια λύση αλλά άμα πάω έρθω σε εσά ή πάω στον κύριο Χουντή θα μου πει όχι δεν θέλω εγκατάσταση καύσης στην Ελλάδα δεν είναι καλό για το περιβάλλον λοιπόν εδώ προ, πρόκειται για θέματα τα οποία δεν είναι μόνο αρμοδιότητο τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Εδώ εμπλέκεται και η περιφερειακή ανάπτυξη. Ε, έχουν οριστεί κάποια κονδύλια για κάποιε με ανοιχτέ εγκαταστάσει που θα κάνει, μηχανική, θα ε, διαλογή, ανακύκλωση κλπ. Και Αυτά όλα θα γίνουν ε, ε, ε, περιμένοντας να φτάσουμε στο τελικά αποτέλεσμα. please. Thank you. Ευχαριστώ. Αφού άκουσα όλες τις παρεμβάσεις, μπορώ να πω ότι δεν πληροφορηθήκα ορθά. Γιατί ακούω αντιφατικές παρεμβάσεις. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν, μας είπατε ότι έγινε μια κρόαση σε δικαστήριο το Μάρτιο σε ένα το δικαστήριο και εγώ είμαι με από τους τέσσερις βουλευτές που θα μεταβούν στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει με απόφαση από το δικαστήριο. Εγώ πραγματικά σας έχασα. Θα υπάρχει μια πραγματική απόφαση από εγχώριο δικαστήριο το θέμα ή όχι. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και αν λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν μπορούμε ριζικά να αλλάξουμε την κατάσταση, Δηλαδή, εσείς ε, από ό,τι κατάλαβα είπατε ότι δεν υπήρχε παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα κατά την άποψή σας. Και απλώ πρέπει να περιμένουμε το 2020 να περιμένουμε 7 χρόνια για να δούμε αν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Εγώ δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη η υποστολή μας. Νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τις διαδικασίες. Αν εσείς δεν πιστεύετε κάτι τέτοιο, θα ήθελα να μου εκφράσετε περαιτέρω επιχειρήματα. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτά. Ε, Γκουράκη, επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, ακούγοντας τους εκπροσώπους της ε, Επιτροπής, οι ανησυχίες μου γίνανε ακόμα πιο μεγάλες. Και θα σας πω γιατί. Οι, οι και οι, οι εντάσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή στο θέμα του ερωτήματος αν η χωροθέτηση είναι σωστή, ή όχι, δεν ακούσαμε καμία απάντηση από τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Και σε άλλα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που ε, έθεσε ο κύριος Γκίκας. Το δεύτερο. Θα ήθελα να σημειώσω λίγο, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν μπορεί σε αυτή την αίθουσα να χρησιμοποιείτε το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα κανεί δεν θέλει χωματερή και άρα κάπου τέλο πάντων πρέπει να πάει. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και επί των συγκεκριμένων πραγμάτων πρέπει να δοθεί και μια απάντηση. Και ε, οι κυρίε τη Κομισιόν ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε μια χώρα με μια, με μια φοβερή υποβαθμισμένη ποιότητα ζωή, λογικό είναι βεβαίω οι κάτοικοι να μην θέλουν μέσα στα πόδια τους να έχουν ε, εγκαταστάσεις τέτοιες οι οποίες θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο το μέλλον και ειδικά το γραμματικό. Ξέρουμε ότι είναι εκτεθειμένο και σε πυρκαγιές, είναι ε, εκτεθειμένο σε καταβληστήσεις, σε μια σειρά από τέτοια ε, φαινόμενα. Και τέλος, εντάξει, υπάρχουν μελέτε άκουσα εδώ μελέτη του Πολυτεχνείου, δεν ξέρω ποια άλλη μελέτη, αλλά υπάρχει ένα θέμα γιατί δεν πείθονται. Δεν πείθονται ούτε οι κάτοικοι, ούτε οι δήμαρχοι, κανένα, Που νομίζω ότι έχουν δίκιο και ακριβώ επειδή ε, δεν άκουσαμε συγκεκριμένη τοποθέτηση για τις συγκεκριμένες ε, ε, αιτιάσεις όσον αφορά ποια είναι η αρχή που έδωσε την άδεια. Εάν είναι ρέμα δεν είναι ρέμα, νομίζω ότι έχουν δίκιο κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σε απάντηση στον κύριο Κουνινιώτη όσο αφορά ότι δεν γνωρίζει τι θα διαχειρίζονται στο, όσο αφορά στο χιτά τον ενημερώνω ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων διαχείρισης για το γραμματικό είναι ένα κδάι 72.000 τόνων ανά μία μονάδα κομπόστ 40.000 τόνων, ε, ένα εργοστάσιο βιολογικής ξύρας CRF δυναμικότητας 127.000 τόνων και οχητά ε, διάθεσης 127.000 τόνους. Ε, άκουσα τον κύριο Κρεμλή. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Κρεμλής λέει τους, τους Έλληνες ανόητους. Δεν μπορούν να κάνουν ανακύκλωση εγώ αυτά κατάλαβα. Ε, θα, θα, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κελμή τι θα κάνει το CRF από τα τέσσερα εργοστάσια. Γιατί το συνολικό, συνολικό ποσό CRF που πρόκειται να κατασκευαστεί α, και από τα τέσσερα εργοστάσια ε, το ξεπερνάμε όλοι σαν ε, η Ελλάδα, το ξεπερνάει από όλη την Ευρώπη. Και όσον αφορά για τον κύριο Κουνινιώτη, μέχρι τώρα μελέτες πανεπιστημίων που έχουμε ε, καταθέσει, έδρες πανεπιστημίων, όχι από τρεις καθηγητές που είναι αυτή η μελέτη, εργαστήρια, ναι, αλλά ε, συγγνώμη, Democracy University, Department of Environmental Engineering, Professor Dr. Ραψομανίκης. Έδρα δεν είναι. Τομέας. Πολύ ωραία, συγγνώμη για το λάθος, τομέας Υπάρχει διαφορά. Τομέα. Ναι, αλλά οι τρει καθηγητέ που υπογράφουν στο MEP ε, ε, είναι τρει. Δεν είναι ο τομέα ε, του συγκεκριμένου του Πολυτεχνείου. αυτή πώ τη δέχεται και την αναφέρει και δεν αναφέρει τι πανεπιστημιακέ μελέτε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου του κ. Κελεπετζή και την, του κ. Ραψομανίκη. Τα αποτελέσματα τα είδαμε στο Καργουνάρι. Μέχρι τώρα, και ο κ. Παπαδόπουλο θα ήταν καλό ένα λεπτό να μιλήσει, αν του δώσετε το λόγο. Ε, τα αποτελέσματα είδαμε. Ο, η, η Επιτροπή είχε πάρει ε, υπέρ το μέρος της, α, α, των ελληνικών αρχών. Μέχρι τώρα είδαν πρόδειλα σφάλματα. Υπάρχει μόλυνση. Ο νομάρχης εκεί, ο περιφερειάρχης που έδωσε τη λειτουργία του Χιτάσου Καρβουνάρη καταδικάστηκε για δεν ξέρω τι ακριβώς. Ε, έχει κατα... διαφθορά γιατί ε, με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεχόταν. Εν πάση περιπτώσει, η διαφθορά είναι μεγάλη. Ευχαριστώ η διαφθορά δεν συμβάλλει στην ερώτηση που μας αφορά εδώ, αφορά εμάς και την Ελλάδα. Παρακαλώ, εδώ πρέπει να έχουμε τα δεδομένα για να δούμε αν υπάρχουν παραβάσεις ουσιαστικές. Ωραία. Ε, δεν ε, αντιλέγω, αλλά πρέπει να βρεθούν. Κύριε φαταλιτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς ε, Εγώ είμαι φίλος της ε, Ελλάδας, είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ την Ελλάδα, σχεδόν όσο αγαπώ και τη χώρα μου. Να κάνω κάποια σχόλια. Είναι προφανώς, ε, είναι προφανές ότι ε, και στην Ελλάδα, όπως και στην περίπτωση της χώρας μου, στη Ρουμανία, δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, τη συλλογική διαχείριση των απορριμμάτων. Όμως κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε κανείς από την Ελλάδα δεν φαίνεται να ανησυχεί γι' αυτό. Επίσης, είναι προφανώς ότι ακόμη και αν η Κομισιόν φαίνεται να έχει μια στρατηγική για την αύξηση του ποσοστού των αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, ε, μεταξύ άλλων. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτή η στρατηγική αφήνεται εντελώς κατά μέρου, σχεδόν εντελώ κατά μέρου και δεν εφαρμόζεται. Ίσως ε, η Κομισιόν να πιστεύει ότι είναι άδικη αυτή η δήλωση, αλλά δείτε ε, τις εικόνες που μας παρουσίασαν εδώ οι αναφέροντες είδαμε συστηματική και κατάφορη παραβίαση των εθνικής, εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα τελήματα σε μία ε, χωματερή, σε ένα χώρο τέτοιο βλέπουμε τα αρέματα να περνάνε ε, μέσα από τα απορρίμματα και η Κομισιόν ε, δεν βλέπει κανένα πρόβλημα εκεί με το σεβασμό και τη, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, και με τα πρότυπα ανακύκλωσης. Τι άλλο μπορώ να πω πέρα από ότι πρόκειται για ε, πρόδειλη καταπάτηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όταν ε, βλέπω να κινείται το έδαφος και όταν βλέπουμε να έχουμε εδάφη που δεν είναι ασφαλή, που είναι ασταθή, αλλά επιτρέπεται παρόλα αυτά να κατασκευαστεί και μια τέτοια κατάσταση. Δεν ε, επιβλήθησαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρξαν κανένα μέτρο διόρθωσης, ούτε καμία κίνηση να αλλάξει η κατάσταση από τις ελληνικές αρχές. Αφού παρακολούθησα αυτές τις δραματικές εικόνες, συμπεραίνω το εξή. Είναι τουριστική χώρα η Ελλάδα και ο τουρισμός ε, είναι πραγματικά ένας μεγάλος πλούτος ε, και θα έπρεπε η Ελλάδα να υπερασπίζει το περιβάλλον γιατί ε, πρέπει να προστατεύσει αυτό το θησαυρό και να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Όμως τέτοιες καταστάσεις οδηγούν σε τρομερές εικόνες όπως αυτές που μόλις είδαμε. Έχω ένα πολύ απλό για την Κομισιόν. Εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια Μιλάμε για ευρωπαϊκά πρότυπα, περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων που δεν γίνονται σεβαστά. Και η Κομισιόν ε, μας ε, δίνει κάποιες απαντήσεις εξ ουρανού, σύμφωνα με τις οποίες η πραγματικότητα που βλέπουν στην Ελλάδα είναι διαφορετική από αυτό που αντιλαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Και κάποιος είπε ότι ίσως ε, θα πρέπει ε, να φεύγουν τα απορρίμματα από την Αττική. Συζητήθηκε στην ε, Αλβανία να απαγορευτούν οι εισαγωγές αποβλήτων, ενώ στην ε, Ρουμανία βλέπουμε τέτοιες εισαγωγές αποβλήτων, πολλές φορές γίνεται αυτό παράνομα και προέρχονται τα απορρίμματα από την Ιταλία και από άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν θέλω να παροτρύνω την Κομισιό να κάνει τη δουλειά της, είστε υπεύθυνοι γι' αυτό και και η πρωτοβουλία του κυρίου και η έκθεση του κυρίου Χουντή αλλά και άλλες δικές μας πρωτοβουλίες πρέπει να σταματήσουν αυτή την αλυσίδα παρατυπιών. Είναι σίγουρο ότι θα μάθουμε πολλά περισσότερα από την ε, αποστολή στην, τις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα. κύριε Κρεμίλια, αν έχετε κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ναι. Θα ήθελα να διασφαλίσω τον Ευρωβουλευτή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τη δουλειά της και βεβαίως υπάρχει σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα. Κάποιες εγκαταστάσεις πρέπει να αναθεωρηθούν βεβαίως λόγω της νέας οδηγίας. Για την Αττική έγιναν ορισμένα πράγματα βάση της οδηγίας του 2003 που αναθεωρήθηκε έκτοτε το σχέδιο να, ε, εγκρίθηκε από όλες τις κυβερνήσεις και επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν βεβαίως ε, πολλές προσφυγές στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα γιατί είναι εύκολη πρόσβαση, οποιοδήποτε μπορεί να προσφύγει. Ε, εγώ όμως θα ήθελα να τονίσω ότι ο, ο δικαστής που εφαρμόζει το ευρωπαϊκό δίκαιο σε τελευταία ανάλυση είναι ο εθνικός δικαστής. Βεβαίως υπάρχει προσφυγή στο δικαστήριο και έχουν επιβληθεί πρόστιμα για τις χωματερές στην Ελλάδα εμείς εκείνο το οποίο τώρα επιμένουμε για την Ελλάδα είναι ότι ε, χρειάζεται να κάνουμε καταστάσεις για τα απόβλητα υψηλότερης αν θέλετε απόδοσης και πάνω από το να είναι απλές χωματερές. Η Ελλάδα λέει ότι έχει το χώρο, μπορεί να ε, έχει απλές χωματερές κτλ. Λοιπόν, προς το παρόν δεν έχει ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ. Οι διαγωνισμοί, είναι εκεί, οι προκηρύξεις βρίσκονται εδώ, δεν έχουν οριστεί ακόμη οι τα ποσά, ούτε οι ποσότητες, ούτε οι τεχνολογίες που θα επεξεργασίας αποβλήτων θα χρησιμοποιηθώ. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Γκίκα δεν είναι CRF, είναι SRF. Δεν πρόκειται να παράγουμε ε, SRF. Κατά πάσα πιθανότητα θα παράγουν RDF. Το θέμα είναι τώρα πώς θα γίνει η διαχείριση του RDF. Έτσι. Και εδώ πρόκειται για το RDF τι είναι, είναι ένα δευτερογενές καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται τσιμεντοβιομηχανίες και τα λοιπά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα τα πούμε μετά το γραμματικό, επομένως μέχρι τότε μένει σίγουρα ανοιχτή, ε, ίσως και αργότερα η ε, καταγγελία ή αναφορά. Παρακαλώ τον κύριο Τούσα για το επόμενο θέμα, ανάλογο. Το πρόβλημα στο γραμματικό δεν είναι ε, ξεχωριστό σε ό,τι αφορά με το ζήτημα που απασχολεί τους χιλιάδες κατοίκους ε, στο Δήμο Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Είναι ο κανόνας για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά και στην προστασία του περιβάλλοντος ε, στην Ελλάδα. Τι θέλουμε να επισημάνουμε. Η αντιλαϊκή πολιτική της ε, τρικοματικής κυβέρνησης στη χώρα μας, Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ρημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτυπάει άγρια τα δικαιώματα των εργαζόμενων αλλά έχει και σοβαρές επιπτώσεις, καταστρέφει το περιβάλλον, βάζει σε τεράστιους κινδύνους τη δημόσια υγεία, την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έκφρασης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής είναι τα μεγάλα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κάτοικοι στο Δήμο Ερμιονίδας, Αργολίδας, της περιφέρειας Πελοποννήσου τα προβλήματα των εργαζομένων κατοίκων της περιοχής έχουν προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Και πώς τεκμηριώνεται αυτό σε σχέση με την τελευταία συζήτηση πριν 1,5-2 χρόνια στην Επιτροπή σας. Από τα επίσημα στοιχεία και τις επιστημονικές αναλύσεις που είναι αναρτημένες τόσο στο Δήμο Ερμιονίδας αλλά και στα σχετικά έγγραφα των αντίστοιχων Υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτο, τεράστιες είναι οι λήψεις στις δημόσιες υποδομές παροχής νερού για ίδρυυση και άρδευση. Ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αν κάποιος ανατρέξει στο διαδίκτυο στη δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης του Τίμιου Ερμιονίδας στην ανακοίνωσή της στις 20 του Μάρτη του 2013 θα διαπιστώσει ότι τεκμηριωμένα το πόσιμο, το νερό του Δήμου Ερμιονίδας είναι ακατάλληλο. Κυβέρνηση και τοπική διοίκηση αντί να πάρουν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος αδειοδοτούν τουριστικά έργα επιχειρηματικών ομήλων, όπως είναι η εταιρεία Might Compass, και ενώ εδώ διψάει η περιοχή πάνω από 16.000 εργαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής, η τοπική διοίκηση του Δήμου Ορμηνίδας, η πλειοψηφία της και η περιφερειακή διοίκηση της Ανατολικής Πελοποννήσου, αντί να προσπαθήσουν να επιλύσουν έστω να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους και τους κατοίκους προστρέχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της εταιρείας Mind Compass για την ε, κατασκευή τουριστική ε, τουριστικής μονάδας με γήπεδο γκολφ, υδροβόρα δραστηριότητα που περιλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης στον κόλπο της Κοιλάδας και θα αποτελέσει τη χαριστική βολή για το περιβάλλον στην περιοχή που είναι ήδη επιβαρημένο. Δεύτερο, έχουμε ετοιμάσει ένα σύντομο τέσσερα λεπτά ε, βίντεο να δείτε τις εξελίξεις ό,τι αφορά ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή. Οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της περιοχής πήραν την υπόθεση στα χέρια τους και όπως βλέπετε απάνω στο βίντεο γολ πάνω από 45.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν συσσωρευτεί στην περιοχή Σταυρός Κλάδεμα στο τοπικό διαμέρισμα διδήμων του Δήμου Ερμιονίδας. Πήραν την υπόθεση ήδη οι εργαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής και έκλεισαν αυτόν, τον άθλιο, αυτή την άθλια κατάσταση που βλέπετε ήδη στο δεύτερο επάνω. Ανοιχτές χωματερές και τάφροι υπάρχουν στην περιοχή όπου θα ε, θάβονται χωρίς κανένα έλεγχο στερεά απόβλητα από την επεξεργασία στην κατεφημισμό αποκαλούμενη μονάδα βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων που βρίσκεται στον κάμπο του κρανιδίου του Δήμιου Ερμιονίδας. Η καθήλια αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης περιφερειακής διοίκησης της περιφέρειας Πελοποννήσου σε έλεγχο που έχει κάνει τεκμηριωμένα έχει διαπιστώσει ότι αυτή η μονάδα δεν λειτουργεί με βάση του ισχύοντες κανόνες και την γενικότερη νομοθεσία. Ε, είναι σοβαρό το ζήτημα ακόμα που υπάρχει σε ό,τι αφορά με την ανεξέλεκτη λειτουργία ιχθυοκαλλιεργιών στον κόλπο, στον αργολικό κόλπο, όπου ενώ οι ίδιες οι αρμόδιες περιφερειακές και υπηρεσίες έχουν εκτιμήσει ότι είναι πολλαπλάσια πλέον η έκταση που καλύπτουν αυτές οι επιχειρήσεις, δεν παίρνουν κανέναν έλεγχο σε ό,τι αφορά για την ποιότητα και το μέγεθος της παραγωγής. Είδαμε από το πρόγραμμα ότι προτίθεται η Επιτροπή το επόμενο χρονικό διάστημα να επισκεφτεί ε, την Ελλάδα και το Δήμο Ερμιονίδας. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να σας μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών, των αλλιέων, των μικρών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ότι η κατάσταση στην περιοχή έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Και πού βλέπουμε εμείς την ευθύνη εδώ και της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές. Με την συγκάλυψη και συνενοχή τόσο της πλειοψηφίας της τοπικής διοίκησης του Δήμιου Ερμηνίδας αλλά και της περιφέρειας με την κεντρική κυβέρνηση αυτό που θέλουν να βάλουν στο χέρι επιχειρηματική ομιλή που δραστηριοποιείται εκεί είναι τα κονδύλια, τα κοινοτικά και κρατικά, έτσι ώστε χωρίς κανένα κόστος να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους σε βάρος τη ε, της ζωής τη ποιότητα ζωή των κατοίκων Ευχαριστώ. σε βάρο του περιβάλλοντο. Τελειώνετε κύριε Τούστα, παρακαλώ. Ναι, θα τελειώσω κυρία Πρόεδρο, αλλά να πω το εξή πράγμα. Παρακολούθησα και προηγούμενα τη συζήτηση. Ε, δόθηκε όλο ο απαιτούμενο χρόνο ε, στου ε, ομιλητέ. Με τα εξή ζητήματα που κατά την άποψή μα είναι γνωστό ότι δεν μπορείτε ως Επιτροπή να δώσετε άμεση λύση σε αυτά Παρά όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία διεκδικούν και παλεύουν οι εργαζόμενοι της περιοχής και είναι το εξής. Πρώτο, να εξασφαλιστεί φθηνό υγιεινό νερό για το Δήμο Ερμιονίδας, αποκλειστικά από δημόσιο φορέα, με την αξιοποίηση των πηγών του Ανάβαλου και του φράγματος ρόλου Τζατζελιάς της Αργολίδας. Το νερό, ο πολυτιμότερος φυσικός πόρος, πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Δεύτερο, να μεταφερθούν τα απορρίμματα σε ασφαλείς χώρους εξεργασίας, να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας στο Σταυρό Κλάδεμα των Διδήμων, του Δήμου Ερμενίδας της Αργολίδας και να αποκατασταθεί το περιβάλλον στην περιοχή. Τρίτο, να διαμορφωθεί αποκλειστικά δημόσιος ενιαίας φορέας διαχείρισης απορριμμάτων με ευθύνη του κράτους και της τοπικής διοίκησης. Τέταρτο, να γίνει έλεγχος της εγκαταστάσει και τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασία αστικών λιμάτων στον κάπο του Κανιδίου του Δήμου Ερμηνεωνίδα. Πέμπτο, να ελεγχθούν οι χτιοκαλλιέργειε και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του αργολικού κόλπου και έκτο τέλος να προστατευτούν τα αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής, το σπήλαιο Φράνθη και άλλα που αποτελεί όχι μόνο πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Τούσα. Ο κύριος Κουνιώτης από την Επιτροπή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο <clears throat> για να μην σα καθυστερήσω κιόλα. Ε, Όπω είχαμε ενημερώσει στην Επιτροπή σα ε, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφασίσει να ανοίξει φάκελο παραβίαση με στοιχεία 2012-2184 κατά της Ελληνική δημοκρατίας λόγω ελλειπής λειτουργίας της εγκατάστασης <clears throat> επεξεργασίας αστικών λιμάτων λιμάτων Ιωνίδας. Η προειδοποιητική επιστολή που επέστειλε η Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2012 αφορούσε ως εκ τούτου την παραβίαση της οδηγίας 91-271 για τα αστικά λίματα. Θα ήθελα να διευκρινίσω, ε, καταρχήν να, να, μιλήσω για δύο άλλα θέματα. Ε, τον Απρίλιο του 2012 είχαμε ενημερώσει την Επιτροπή σα για του λόγου για του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμάει ότι δεν υφίσταται πλέον παραβίαση τη Οδηγία 9883 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινη κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική δημοκρατία είχε λάβει βάση του άρθρου 8 τη οδηγία αυτή τι αναγκαίε επανορθωτικέ ενέργειε για την αποκατάσταση τη ποιότητα του νερού στο Δήμο ενώ παράλληλα και για τη μεταβατική περίοδο μέχρι να, να τεθούν σε λειτουργία αυτέ οι ενέργειε, είχε θεσπίσει σύστημα παρακολούθηση τη ποιότητα του νερού και σύστημα ενημέρωση των καταναλωτών. Για το δεύτερο θέμα που, κύριε, που μιλήσαμε προηγουμένως για τον Χαδά ε, Σταυρού Κλάδεμα, η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα αυτό. Είναι εξάρου μία από τις ανεξάρτητες χωματερές που συμπεριλαμβάνονται στην υπόθεση για την οποία η Επιτροπή προσέφυγε το Φεβρουάριο του 2013 στο, στο δικαστήριο για δεύτερη φορά ζητώντας ε, καταβολή προστίμου. Ε, εδώ απλώς θα επαναλάβω ότι ε, η Επιτροπή βέβαια θα, ε, απαιτεί το κλείσιμο του Χαδά και την αποκαταστασή του, αλλά αντικειμενικά για να γίνει αυτό τα σκουπίδια που μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στο Χαδά θα πρέπει να μεταφέρονται σε μια κατάσταση που πρέπει να δημιουργηθεί. Ε, λοιπόν, για να επανέλθω τώρα στην προοδοποιητική επιστολή και στα αστικά λήματα, ε, οι ελληνικέ αρχέ μα έχουν απαντήσει και παρά το γεγονό ότι δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρω με την οδηγία, ε, παρατηρούνται ε, ε, μία μερική πρόοδο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, παρά το γεγονό ότι μόνο ένα 20% του οικισμού του κρανιδίου εξυπηρετείται από το αποχετευτικό δίκτυο, τα υπόλοιπα αστικά λύματα αποχετεύονται εμέσως προς την υπάρχουσα εγκατάσταση επεξεργασίας μέσω της μεταφοράς βοθρολυμάτων προς προσωνή δεξαμενή. Κάτι τέτοιο ε, εξάλλου επιτρέπεται από την οδηγία στο άρθρο 3, εφόσον βέβαια, και το τονίζω, επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, το ίδιο επίπεδο. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ενώ στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί διαρροές και μόλυνση του περιβάλλοντος, αυτή η νέα δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και βρίσκεται πλέον εντός του κλειστού και φυλασσόμενου χώρου της εγκατάστασης. Δηλαδή η ανοιχτή χωματερή δεξαμενή που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν έχει πλέον σταματήσει να χρησιμεύεται και δεν υπάρχουν ελλείμματα. Άρα δεν υπάρχουν και διαρροές. Δεύτερον, το σύστημα χλωρίαση τη εγκατάσταση λειτουργεί Τρίτον, καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας της μονάδας και συντόμως αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι υπάρχουσες εφεδρικές δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης, οι οποίες ουδέποτε μέχρι τώρα λειτουργούσαν. Τέταρτον και τελευταίο, οι μελέτες του έργου αποπεράτωσης αποχαιρευτικών δικτύων κρανιδίου, αγωγή μεταφοράς λιμάτων και μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολιμάτων έχουν πλέον επικαιροποιηθεί και έχει υποβληθεί αίτημα για την χρηματοδότηση του έργου στο αρμόδιο Υπουργείο. Η λειτουργία του έργου αυτού θα εξαλείψει τα προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος που παρατηρούνται μέχρι και σήμερα, ενώ θα μειώσει και το κόστος λειτουργίας της μονάδας. Βέβαια, παρά αυτέ τι θετικέ εξελίξει, η μονάδα δεν πληρεί ακόμη τι απαιτήσει τη οδηγία για τα αστικά λίματα, όπω εξάλλου φαίνεται και από την τελευταία ε, αυτοψία που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Και ένα τελευταίο σημείο, δεν υπάρχουν ακόμη εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση. Για αυτού του λόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να επιτηρεί την κατάσταση και αν δεν επιτευχθεί σύντομα πλήρη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών, δεν θα διστάσει να αποχωρήσει στο επόμενο στάδιο και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Αγκουράκη. Ευχαριστώ, κυρία... Πρόεδρε. Ε, νομίζω από την ε, αναφορά ε, φαίνεται ένα σύνολο προβλημάτων που, που απασχολεί τους ε, κατοίκους της περιοχής και δικαιολογημένες είναι αντιδράσεις και διαμαρτυρίες τους. Φαντάζομαι ότι με την επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας της Επιτροπής και επιτόπου θα διαπιστώσετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Φαίνεται ότι στο βασικό πρόβλημα, το, ένα από τα βασικά προβλήματα που είναι το πρόβλημα του νερού, είναι απόλυτα τεκμηριωμένες και απόλυτα επιβεβαιωμένες οι διαπιστώσεις και οι καταγγελίες ε, μάλιστα θα ήθελα να πω κύριε ε, κυρία Πρόεδρε ότι και από την απάντηση της Κομισιόν ε, οι ανησυχίες μου ενισχύθηκαν διότι τι, τι απάντηση πήραμε πήραμε ότι έχει, έχει εγκατασταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος ελέγχει την ποιότητα του νερού και προειδοποιεί τους κατοίκους. Δεν πήραμε την απάντηση ότι η ποιότητα του νερού είναι αυτή που πρέπει να είναι και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ε, επίσης, ε, καμία τοποθέτηση δεν ακούσαμε για το θέμα του εργοστασίου αφαλάτωση, που προφανώς θα έχει σοβαρέ επιπτώσεις ε, στην περιοχή και στο περιβάλλον, όπως επίσης τίποτα για το θέμα των ηχθιοκαλλιεργειών, που δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμες, είναι παράνομες, τηρούν τις προδιαγραφές ή όχι. Για τα αρχαιολογικά δεν επεκτείνουμε, εδώ φαίνεται δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό το ζήτημα Ειδικά εσά όμω σα ενδιαφέρει ιδιαίτερως από ό,τι ξέρω και όλου του ε, υπόλοιπου. Για να καταλήξω στο εξή. Ε, αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται ε, συμπίεση των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπίεση των απολαβών των εργαζομένων, αυτή η επίθεση στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, είναι προφανέ ότι έχει πολύ σοβαρέ επιπτώσει και στα πολύ σοβαρά προβλήματα και ζητήματα που καταγγέλνουν οι κάτοικοι τη Ερμιονίδα. Και δυστυχώς επειδή αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί και θα ενταθεί στο άμεσο μέλλον ε, για πολλούς και διάφορους λόγους που γνωρίζουμε και κυρίως για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, ανησυχούμε πάρα πάρα πολύ και για τις καταγγελίες που έχουν σχέση με την ε, ανάπτυξη τουριστικής μονάδας στην περιοχή. Ξέρετε, στο όνομα του, του κέρδους και των επενδύσεων πολλές φορές έχουν παραβιαστεί και έχουν παραμεληθεί στοιχειώδεις ε, έργα και στοιχειώδεις υποχρεώσεις και γι' αυτό το λόγο είμαστε πραγματικά στο πλευρό των, των κατοίκων. Μαζί του θα αγωνιστούμε τουλάχιστον ορισμένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπιστούν και να παρθούν τα μέτρα όπω θα προτείνουν εκείνοι, ώστε, γιατί είναι και συγκεκριμένε οι προτάσει που κάνουν, δεν είναι δηλαδή ευχολόγια, ώστε να διασφαλιστεί ένα ανεκτό επίπεδο ε, ζωή. Ευχαριστώ. Και για έχετε καταθέσει στη Γραμματεία ε, Είναι προτάσει που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα επανέλθουν. Αλλά αν δεν υπάρχει άλλο συνάδελφο. Επίση. Απευθύνομαι προ εσά, στου ευρωβουλευτέ. Απευθύνομαι προ τον Πρόεδρο, του ευρωβουλευτέ και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί παίρνετε μια πολύ τεράστια μεγάλη ευθύνη να συγκαλύψετε και έχω συνέστηση αυτό που λέω και θα σας το αποδείξω ένα έγκλημα που είναι σε εξέλιξη σε βάρος των εργαζόμενων των κατοίκων της περιοχής. Το πρωί από το διαδίκτυο είναι στη διάθεσή σας. Είναι οι αναρτημένες αναλύσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού στο Δήμο Ερμιονίδας όπου υπάρχουν περιπτώσεις που είναι οι δείχτες των συστατικών στοιχείων όπου ξεπερνούν τα όρια που καθορίζονται σε ό,τι αφορά την κοινή υπουργική απόφαση και τα κριτήρια είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους ότι το νερό δεν χρησιμοποιείται για πόσιμο. Πάει πολύ λοιπόν να έχωσαστε παρουσία σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών και να λέτε ψέματα. Όχι, ε, όχι, όχι. Ε, εμείς, καταθέτουμε τα, χαρτιά, εμείς καταθέτουμε τα χαρτιά, είναι, θα τα καταθέσουμε εσάς, λέτε ψέματα. Και ε, παραπλανάτε και τους ευρωβουλευτές αλλά και τα κριτήρια της αξιολόγησης. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ε, δεν μπορεί να μείνει έτσι. κύριε Τούσα να πάρετε πίσω το λέτε ψέματα. Καθόλου, Έχω συνέστηση, Ωραία. έχω πάρα πολύ μεγάλη Ωραία. συνέστηση και η συνέστησή μου αυτή είναι ότι ε, η υγεία, με την υγεία χιλιάδων εργαζόμενων κατοίκων της περιοχής δεν μπορεί να παίζει κανένας. Αν σήμερα βγήκα στο διαδίκτυο, γιατί... Όχι, από 20 του Μάρτη. Να προχωρήσουμε. Θέλετε κάτι να πείτε κύριε Κουνινιώτη. Απλώς... Ε, όχι απλώ για, για, τα λέτε ψέματα. Ε, δεν ξέρω πώ δεν είναι καλά κατανοητό. Ε, όσο αφορά την ποιότητα του ανθρώπινου νερού, δεν είπαμε ποτέ ότι είναι καλή. Είπαμε ότι λαμβάνονται ε, μέτρα. Οπότε. Κοιτάξτε, δεν τα έχω κατα... μπροστά μου εδώ πέρα όλη τη λίστα, δεν είμαι σε θέση. Οπότε, αν, αν, αν υπάρχουν μέτρα τέτοια, σημαίνει ότι η ποιότητα δεν είναι καλή. Γι' αυτό και λαμβάνονται μέτρα. Οπότε δεν βλέπω γιατί είμαστε ψεύτες που λέμε ότι λαμβάνονται μέτρα. Ευχαριστώ. Πέστε μας τα μέτρα, τα μέτρα. Πέστε μας ένα Ζητήστε το στο κοινοβούλιο το ελληνικό. Δεν το έχω πέσει. Ε, ε πρώτα, απ' όλα το μέτρο. Πρώτα απ' όλο. Ναι. Το, το μέτρο, το πρώτο μέτρο. Το είναι υπο... Sorry, Madam Chair, but this is not a Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, εδώ δεν είναι μαχοπέδιο Μα... για καυγάδες μεταξύ των Ελλήνων της Κομισιόν και των Ελλήνων της Ελλάδας ή του Κοινοβουλίου. Συγγνώμη, πρέπει να γίνονται σεβαστά και ορισμένα πράγματα, υπάρχουν όρια. Let's go to the next petition. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου για την παρέμβασή σα. Ε, φυσικά αυτή, αυτή η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή. Α πάμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε την αναφορά του Ιαντρέα Ρουτιλιανού από την Ιταλία. Όχι. Το υπερθυμό 12. Καταρχήν για τη Βάγια Γκαλέρια. Ο κ. Ραντόλφο είναι ο Αναφέρον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας διαβάσω την αναφορά μου. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Ροντόλφο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω αυτήν την Επιτροπή για την ευαισθησία που έχει επιδείξει απέναντι στο πρόβλημά μας και συγκεκριμένα ε, να ευχαριστήσω την κυρία Ματσόνη που ε, δέχτηκε με ένα απλό mail την ε, αναφορά μου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτε μου για την οικονομική προσπάθεια και για το χρόνο που, κατε... που αφιέρωσαν ε, έτσι έστω εγώ και ο... έτσι ώστε σήμερα εγώ και ο Πέτρο να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε εδώ τι συμβαίνει με τα απόβλητα ε, στην κοιλάδα γκαλέρια και να σας παρουσιάσουμε τι συμβαίνει με, την, με τα απορρίμματα στην περιοχή. Ήδη υπάρχει μόλυνση λόγω της χωματερής ε, της Μαλαγκρότα, λόγω της εγκατάστασης αποτέφρωσης ε, νοσοκομιακών οχημάτων και λόγω του δηληστηρίου. Η πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό το ταξίδι ε, εκπροσωπεί σε αυτή την πρωτοβουλία έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους όλοι οι πολίτες της Κοιλάδας ε, δεν είμαι εμπειρογνώμονας, όμως θα μιλήσω μόνο για τον πόνο μας και τα τεχνικά στοιχεία θα τα παραδώσω στην Προεδρία. Εμείς ε, είμαστε εδώ γιατί έχουμε κουραστεί, δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε αυτά που συμβαίνουν, μας έχουν ε, οδηγήσει σε συναισθηματική και ψυχολογική κούραση. Καθημερινά πρέπει να ζούμε με συνεχείς διαψεύσεις και δηλώσεις που μόνο μας οδηγούν στην απελπισία. Είμαστε συγχυσμένοι, αποπροσανατολισμένοι, εξαντλημένοι. Όμω είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι τέλους και να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να περασπίσουμε το δικαίωμά μα στην υγεία το οποίο γράφεται στο Τελικό Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πιστέψτε με, γι' αυτό αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ψυχραιμία του όταν συνεχώς τον κροϊδεύουν με δηλώσεις ή οχοδερφιστικές ε, δηλώσεις ε, που γίνονται από κάποιους θεσμούς που δεν έχουν εκλεγεί από κανέναν ε, είτε από κάποιους οι οποίοι αποφάσισαν να αναλάβουν τη διαχείριση των αποβλήτων μας. Επίσης θα έλεγα ότι τέτοιες ε, συμπεριφορές ε, δημιουργούν πραγματική δυσαρέσκεια στον πληθυσμό και δεν ξέρω που θα καταλήξουν τα πράγματα. Έχουμε κουραστεί από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ε, από τις χωματερές, τα δηληστήρια, όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην περιοχή μας. Τα γνωρίζετε και εσείς. Είμαστε κουρασμένοι να συνεχίζουν να μας λένε ότι οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και τα υπόλοιπα αποτελούν ευλογία από το Θεό. Έχετε δει με τα μάτια σας τι συμβαίνει στην Κοιλάδα Γκαλέρια, έχετε δει με τα μάτια σας την περιβαλλοντική καταστροφή στο Μόντι Τελορτάτσιο και εσείς ήδη ε, εκφράσατε την αντίθεσή σας στο να δημιουργηθεί η χήτα. Κι όμως ο Επίτροπος Σεπτήλ επέτρεψε μία άδεια στις 27 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους που μπορεί να εκτελεστεί από νομική σκοπιά για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Μόντι Ντελορτάτσο και καλώντας τον ιδιωτικό τομέα να ελέγξει τον εαυτό του. Και είπε μάλιστα ότι πιστεύετε τον ιδιωτικό τομέα. Ο υπουργό ε, κλείνει με τη σειρά του, ε, μας είπε ότι δεν είναι αλήθεια ότι η έγκριση ισχύει και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ως ε, υπουργός να αποσύρει αυτή την άδεια. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο εμείς οι πολίτες ε, βρισκόμαστε κουντουφλώντας στο σκοτάδι, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος έχει την ευθύνη και να ε, προσπαθήσουμε να βγάλουμε πάνω από το κεφάλι μας αυτή τη δαμόκλειο σπάθη. Ε, όμως ε, ο ιδιωτικός τομέας παρόλα αυτά συνεχίζει με τον καθαρισμό της περιμέτρου του χώρου και ο Υπουργός κλείνει ενώ μας είχε διαβεβαιώσει ότι μόνο για 18 μήνες θα λειτουργούσε η χωματερή. Τώρα φαίνεται ότι θα διαρκέσει ε, η λειτουργία για 36 μήνες. Η, σε όλο αυτό το χάος ε, δεν ε, έχει γίνει μια ορθή περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου και ξέρετε ότι κανονικά αν υλοποιηθεί αυτό ο τότε θα υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις στην Ιταλία πριν ε, λίγες μέρες, αν δεν είχε ε, κλείσει η Μαλαγκρότα, ε, πραγματικά θα βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όμως τώρα βλέπουμε να δημιουργείται μία δεύτερη μαλαγκρότα. Υπαριθμών 2. Κανείς δεν γνώριζε κάτι τέτοιο και δόθηκε η άδεια μέσα σε 24 ώρες από κάποια αρχή που φυσικά εξυπηρέτησε τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά είναι λογικό να αναρωτηθούμε, αλλά από πού ξεφύτρωσε, είχε, ε, ήταν κρυμμένη μέσα σε κάποιο σιρτάρι. Μιλάμε για μια προσωρινή έγκριση, όπως ε, τόσο προσωρινή όσο είναι όλες και αυτό σημαίνει ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 20 χρόνια. Την περασμένη Παρασκευή ένα δικαστήριο ε, θεώρησε ότι ο ιδιωτικό ε, τομέας έχει δίκιο όταν ε, δηλώνει ότι έκανε τις εξκαφές γιατί το 2009 ήδη είχε δηλώσει τις προθέσεις να δημιουργήσει εκεί τη χωματερή. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει ότι μπορεί κάποιος καταχρηστικά να αρχίσει τις καφές. Επομένως, οτιδήποτε αποφασίσει ο ιδιωτικό τομέα εγκρίνεται χωρίς ε, να ρωτήσουν τους πολίτες, χωρίς να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία, για την πανίδα, για την κλωρίδα. Εμείς σε αυτή την κατάσταση ζούμε στη Βαλεγκαλέρια και πέρα από ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε το τέρας της ρήπανση, ε, των χωματερών και των καταστάσεων αποτέφρωσης, πρέπει να ζήσουμε και με ένα χειρότερο τέρας που απειλεί να καταβροχθήσει την αξιοπρέπειά μας. Δεν ξέρουμε πια σε ποιον να στραφούμε για να μας ακούσει. Επομένως, σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε, να μας βοηθήσετε και να ζητήσετε να αποσυρθεί αμέσως η άδεια αυτή, η έγκριση αυτή. Εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε ούτε μία μέρα παραπάνω με αυτόν τον τρόπο, να είμαστε ξεχασμένοι και αποκλεισμένοι από οποιαδήποτε λύση του προβλήματος. Όποιος δεσμεύεται ψυχή και σώματε σε αυτόν τον αγώνα, άφησε κατά μέρου τη ζωή του, τη δουλειά του, τους φίλους, τους δικούς του ανθρώπους. Εμείς θέλουμε μόνο ξανά τη ζωή μας πίσω και την υγεία, τη δική μας και των αγαπημένων μας. Έχουμε κουραστεί να πληρώνουμε τόσο υψηλό μα, επειδή ε, αγαπούμε τη γη όπου κατοικούμε. Σας ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Πίσου παρακαλώ. Για ένα λεπτό μόνο. Καλημέρα σας. Εγώ ζω μια Οδύσσια εδώ και 20 χρόνια. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την δημιουργία αυτής ε, της χωματερής. Και εδώ να συμφωνήσω με τον σύντροφό μου. Θέλω να παρουσιαστώ εδώ σε αυτή την επιτροπή για να σας πω ότι δίκηση μας τον Ιανουαρίο του 2006 έκανε μια αλλαγή ε, χρήσης ε, μιας ε, γης καλλιεργήσιμης για δημόσια χρήση υπήρχαν ε, κάποιες ε, τεράστιες τρύπες ε, γιατί εκεί αφαιρούν υλικά για οικοδομικά. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι η κοιλάδα μας είναι γεμάτη τρύπες και όταν βλέπει κάποιος μια τρύπα πετάει μέσα τα πόβλητα και στη δίκηση μας το επιτρέπουν αυτό. Εγώ όμως δεν θέλω πλέον να συμβαίνει αυτό, είναι αδύνατο. Εμείς αγωνιστούμε μέχρι το τέλος έτσι ώστε να μην συμβαίνει αυτό πλέον. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζητάνογκα. Ζητάνογκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρους της κυρίας Άουκεν, που έλαβε μέρος ε, στην ε, επίσκεψη στην περιοχή που συζητείτε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρούσα. εξήχθησαν θετικά άμεσα αποτελέσματα από εκείνη την επίσκεψη όσον αφορά την αντίδραση των αρχών παραδείγματος χάρη. Αλλά η κυρία Όκεν απογοητεύτηκε από την περαιτέρω αξιολόγηση διότι φαίνεται ότι οι αρχές δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη την επίσκεψη που έγινε και φάνηκε άλλωστε και στον Ιταλικό τύπο ότι τα προβλήματα που αναφέρουν οι αναφέροντες εδώ συνεχίζουν να υπάρχουν. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα από τη μεριά της Επιτροπής ο κύριος Μαγκανάρο. Signore Μαγκανάρο, grazie. Ehm, la questione molto complessa della gestione dei rifiuti nel Lazio è seguita. Oh ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων στο Λάτσιο είναι περίπλοκο. Εδώ και κάμπος εδώ και τρία χρόνια περίπου ε, ε, ασχολούμεθα με συγκεκριμένα θέματα. Βεβαίως υπάρχει κατά παράβαση διαδικασία ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οποία προχωρεί. Η, η εγκατάσταση όμως του Μαλαγκρότα συγγνώμη, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήταν λόγω της ε, ε λειτουργίας της εγκατάστασης στη Μαλακρότα που δεν λειτουργούσε σωστά και άλλα, άλλες εγκαταστάσεις ε, βέβαια δεν γίνεται προεργασία των αποβλήτων και γι' αυτό τα, τα απόβλητα είναι μη σταθερά και δεν συρρυκνώνονται όσο θα έπρεπε έχουν χειρότερες επιδράσεις στο περιβάλλον από ό,τι θα μπορούσαν να έχουν βεβαίως οι Ιταλικές αρχές σκέφτονται να κλείσουν την εγκατάσταση της Μαλαγκρότα ένα άλλο θέμα το οποίο συζητείται και απασχολεί είναι τι θα γίνει όταν οι Ιταλικές αρχές θα ανοίξουν καινούργιες χωματερές ή καινούργια εργοστάσια. Κατά πόσον ακολουθούνται οι διατάξεις των σχετικών οδηγιών, κατά πόσον γίνονται σωστά οι αξιολογήσεις ε, αντικτύπου στο περιβάλλον Μοιραία βεβαίω πριν να ανοίξουν καινούριε εγκαταστάσει κομματερέ θα πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση. Αλλά από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμή στη διάθεσή μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει παράβαση των κανόνων οπότε φαντάζομαι ότι τα σχέδια αυτά θα προχωρήσουν αν όμως τελικά αποδειχθεί ότι υπάρχει παράβαση ορισμένων διατάξεων και η Ευρωπαϊκή τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει καινούργια προσφυγή Κύριε ναι. Κυρία Πρόεδρε, οι αρχαίοι α, Ρωμαίοι έλεγαν «Ράρε ουμάνουμ». Είναι όντως ανθρώπινο το σφάλιν, αλλά και το πότε το εράρε γίνεται περσεβεράρε πότε τελικά θεωρείται ότι έγιναν ορισμένα λάθη ότι έγινε κάποια μελέτη και εξήφισαν τα σωστά συμπεράσματα η Κομισιόν τι κάνει ναι υπάρχουν λάθη, υπάρχουν, πρέπει να γίνουν έλεγχοι, γίνονται. Κλείνει η Μαλαγκρότα, προσφυγή για τη Μαλαγκρότα, προσφυγή δύο για τη Μαλαγκρότα κτλ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα με, Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα, κάθε μήνα μετά από δύο επισκέψεις της Επιτροπής μας στην περιοχή. Μετά από την παρουσίαση στον τύπο όλων αυτών των προβλημάτων στην περιοχή. Πότε η Κομισιόν τελικά θα πει αρκεί, φτάνει πια και θα επιβάλλει ορισμένα πράγματα πότε θα παρθούν αποφάσεις, πότε θα επιβληθούν μέτρα για να σταματήσουν ορισμένα πράγματα. Τώρα με έναν πολύ πλατωνικό τρόπο μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι γίνονται κάποιες απάρθηκαν κάποιες αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο αλλά δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες άπαξ και αρχίσουν οι εργασίες τότε θα αντιδράσουμε Μα τι να αρχίσει. Εδώ και δέκα χρόνια κουβεντιάζουμε τα ίδια πράγματα και καμία κυβέρνηση Ιταλική ούτε από την κεντροαριστερά ούτε από την κεντροδεξιά ούτε η συν, συνασπισμού ούτε μεγάλου συνασπισμού ούτε μικρού συνασπισμού λοιπόν καμία κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους κανόνες και η Κομισιόν ήρεμα και άνετα λέει μόλις παραβιαστούν οι κανόνες εμείς θα δράσουμε ε πως θα δράσετε πότε θα πείτε φτάνει πια που βρίσκεται η διαχωριστή κόκκινη γραμμή Λέω στην Κομισιόν, αυτοί που πληρώνουν τα πρόστιμα είναι οι Ιταλοί φορολογούμενοι. Ο Ιταλικός λαός πληρώνει τα πρόστιμα και πώς θα, βο... επισκευαστεί ή επανορθωθεί η κατάσταση. Η Μαλαγκρότα είναι μια ιστορία 20 ετών. Ταλαιπωρείται ο κόσμος εκεί γύρω. Και δεν αρκεί αυτό. Η Κομισιόν έχει φαίνεται ένα πολύ παράξενο τρόπο να ε, μετράει το πότε το εράρε είναι περσεβεράρε και πότε φτάνει πια Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υπόθεση της Βαλεγκαλέρια είναι μία από τις ε, χιλιάδες ε, ιστορίες που ήδη έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν στην Ιταλία, αλλά και όχι μόνο. Εγώ Μπορώ να σας πω ότι αυτές οι χωματερές και αυτά τα προβλήματα της μόλυνσης των υδροφόρων οριζόντων ε, και των εδαφών είναι φαινόμενα που δεν τα συναντάμε μόνο στην κεντρική και νότια Ιταλία αλλά και στη βόρεια Ιταλία. Εγώ ζω σε μια κοινότητα 22.000 κατοίκων, έχουμε 11 χωματερές ε, και 5 από αυτές ε, τώρα μολύνουν τον υδροφόρο οριζόντα. Στη βρανατολική Ιταλία συνολικά έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο έδαφος ε, γλυκού νερού, αλλά δυστυχώς ε, δεν είναι πόσιμο αυτό το νερό γιατί μολύνεται υδροφόρος ορίζοντες, ε, κυρίως στο παρελθόν μολυνθεί, αλλά και σήμερα και δυστυχώς καταλήγουμε να μην έχουμε πόσιμο νερό. Εγώ νομίζω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να παρακολουθεί εκ του θέμα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Έχουμε την οδηγία για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή του κοινού και μέγιστη διαφάνεια. Υπάρχουν εναλλακτικέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς οι βουλευτές, πέρσι στι 24 Μαου, εγκρίναμε την έκθεση Κάρπαντη για την αποτελεσματική χρήση των πόρων στην Ευρώπη. Σε αυτή την έκθεση λέγεται ότι φτάνουν πια εχομετερές, ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε όλα τα απόβλητα, γιατί είναι πολύτιμο υλικό. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο που δημιουργεί τόσα προβλήματα στο περιβάλλον μας και το ίδιο πρέπει και να το πούμε για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Μέχρι το 2020 πρέπει να δώσουμε τέλος, να θέσουμε τέλος στην καύση των αποβλήτων, πρέπει να μιλάμε για ανάκτηση των αποβλήτων. Έτσι λοιπόν, εμείς στο Βένιτο έχουμε κάποια παραδείγματα αποτελεσματικά και πολύ σημαντικά, όπου Έχουμε πιλωτικά κέντρα στην επαρχία του Τρεβίζο, παραδείγματο χάρη, όπου φτάσαμε σε 100% ανακύκλωση των αποβλήτων, των αστικών αποβλήτων. Επιπρόσθετα, έχουμε διάφορα ε, πάνελ που ήταν αδύνατον να τα ανακυκλώσουμε, ενώ τώρα είναι δυνατόν να γίνει αυτή η ανακύκλωση χάρη σε κάποια συστήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι το 100% αυτών των αποβλήτων. Και κάτι τελευταίο. Αυτή η δραστηριότητα και εμείς ε, απευθύνουμε μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ζητήσαμε, περιμένουμε λοιπόν νομοθετικές προτάσεις, φέρουν και μια οικονομική βοήθεια, κυρίως σε περίοδο κρίσης. Ένα παράδειγμα, χάρη στις πρώτες ύλε που παράγονται από αυτό το κέντρο ανακύκλωσης αποβλήτων, παράγεται, παράγονται κάποια κόκκι πλαστικού έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το ανακυκλωμένο πλαστικό κοστίζει 400 ευρώ ο τόνος. Και αυτή οι κόκκι πλαστικού που δεν είναι ανακυκλωμένοι κοστίζουν 4.000 ευρώ. Ε, το τόνος και στην επαρχία της ε, Φεράρα ε, μία βιομηχανία σώθηκε από το κλείσιμο, ε, γιατί δεν μπορούσε πλέον να ανταγωνιστεί τα κινέζικα προϊόντα, χάρη σε, στην παραγωγή αυτού του ανακυκλωμένου υλικού. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να καταφύγουμε σε τέτοιες λύσεις, ε, να θέσουμε ένα τέλος στη ρήπανση του περιβάλλοντος, να σταματήσουμε την καύση και να χρησιμοποιήσουμε και ε, αυτά τα υλικά που θεωρούμε ότι πρέπει να τα πετάξουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε προς, την, προς ανάκτηση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό στους αναφέροντες, αν ε, έχουν κάτι να σχολιάσουν. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι πολίτη, δεν είμαι εμπειρογνώμονα, αλλά κάναμε κάποιε προτάσει εμεί στη Βαλακαλέρια. Και στην ε, κοινότητα τη ε, Ρώμη, όπου έχουμε τώρα 15 περιφέρειες, ζητήσαμε από το Δήμο τη Ρώμη να χρησιμοποιηθούν κάποιες οικολογικές νήσοι όπου θα γινόταν εκεί η διαχείριση των αποβλήτων. Εμείς έχουμε μόνο μία εγκατάσταση για κόμποστ και δεν αρκεί. Θα χρειαζόμαστε 20 ακόμη αλλά εγώ ως πολίτης πρέπει να πάω στο Δήμο και στους εμπειρογνώμενους και στου πολιτικού να κάνω αυτές τις προτάσεις. Αυτοί πληρώνονται. Αυτοί πρέπει να κάνουν αυτές τις προτάσεις. Εμείς τους έχουμε κλέξει για αυτή τη δουλειά και πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους μέχρι το τέλος. Σα ευχαριστώ και συγγνώμη που τα είπα έτσι έντονα. Υπάρχει ήδη ένα κείμενο που αφορά την επίσκεψη αποστολής στην, τον προηγούμενο χρόνο στην περιοχή. Η άποψη των μελών που την επισκέφτηκαν και εγκρίθηκε από το σύνολο των μελών της Επιτροπής είναι ότι πρέπει να βρεθεί εναλλακτικός χώρος για τα, για τα σκουπίδια. Επομένως, ε, ε, η Κομισιόν γνωρίζει την άποψη της Επιτροπής ε, Αναφορών. Πάμε στην επόμενη αναφορά. Ευχαριστώ όσους ήταν. από την κυρία Σέιλα Έλλης από τη Βρετανία σε σχέση με την αδυναμία της, του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει την οδηγία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Of course the petition was mentioned. The one we are uh, Mrs. Ellis. Thank you. Κυρία Ellis, ευχαριστώ. Καλημέρα σας ε, κυρίες ε, και κύριοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που μας ε, καλέσετε εδώ να αναγνωρίζοντας ότι κάθε άτομο έχει τη δικαίωμα να ζει σε ένα κατάλληλο περιβάλλον για την υγεία του και για την ευημερία του και το καθήκον ε, και ατομικά αλλά και συλλογικά να προστατεύσει και να βελτιώσει το περιβάλλον προς ε, όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενιών θεωρώντας ότι πρέπει να είναι δυνατό να τηρείται και να εφαρμόσετε αυτό το δικαίωμα οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες να συμμετέχουν στη την λήψη αποφάσεων και επίσης ε, να αποδίδεται δικαιοσύνη σε αυτούς σε περιβαλλοντικά ζητήματα και πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να χρειάζονται και βοήθεια οι πολίτες για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ε, αυτό το προήμιο τη σήμερα τη συμπεριλαμβάνεται στο ε, τρένα οι ίδρυτες ε, πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών ε, αναφέρθηκαν στα φυσικά δικαιώματα που, δεν, που είναι ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό, όμως εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια τέτοια αναφέροντα δικαιώματα όπως το οποίο είναι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας. Επομένως, τι θα κάνουμε σαν ένα κράτο μέλος των οποίων τα όργανα της κυβέρνησης συστηματικά ουσιαστικά υποσκάπτουν τα καθήκοντά μας ε, ε, να έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον και τι θα κάνουμε σε ένα κράτο μέλο, τα όργανα της κυβέρνησης συστηματικά υποσκάπτουν ε, τα καθολικά δικαιώματα των πολιτών. Δύο φορές στο παρελθόν έχουμε έρθει εδώ για αναφερθούμε στο τι συμβαίνει στη Βόρεια Αγγλία από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι αρμόδιες ε, να προστατεύουν το περιβάλλον ε, και την υγεία και την ευτυχία των κατοίκων μας αλλά και το καθαρό νερό. Όχι μόνο η τεράστια χωματερή στο μέσο της πόλης μας ε, δηλητηριάζει το νερό και τον αέρα αλλά αυτό έχει αποδειχτεί τώρα και στο δικαστήριο και δυστυχώς οι περιορισμένες διώξεις ε, ε, που έχουν ασκηθεί από την περιβαλλοντική αρχή δεν αρκούν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, πέντε υποθέσεις ε, που ε, συζητήθηκαν στο δικαστήριο γιατί καθημερινά στραγγίδια διαραίουν τα τελευταία 13 χρόνια από τη χωματερή από το Μάιο του 2012 λόγω της ρήπανσης σημαίνονται προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα. Έχει επίσης φανεί ότι είναι σε ε, ε, η χωματερή βρίσκεται πάνω σε σαθρούς βράχους που καταστρέφουν ε, τα συστήματα στεγανοποίησης και παρόλο που είναι παράνομο να παράνομη άδεια που έχει δοθεί η περιβαλλοντική υπηρεσία του Ερμένου Βασιλείου αρνείται να αποσύρει την άδεια και αρνείται να διώξει το φορέα εκμετάλλευσης. Η υπηρεσία μας λέει ότι ποτέ δεν έχει σταματήσει τη λειτουργία της ε, χωματερής ε, και δεν έχει καμία σημασία πόσο κακά έχει κατασκευαστεί και λειτουργήσει και παρόλα τα ψέματα και παρόλο τα δεινά που, έχουν υποστεί οι πολίτες, ποτέ δεν ε, έχουν αποσύρει την άδεια. Οι εκπρόσωποι ε, της ε, χώρας μας εντελώς κοινικά όχι μόνο δεν έχουν σεβαστεί το νόμο στο πνεύμα του, αλλά ούτε στη θεωρία. Ως Ευρωπαίοι πολίτες, εμείς έχουμε παρουσιάσει τεχνικές αποδείξεις για ότι πάνω από 10 χρόνια υπάρχει τεράστια ρήπανση στο περιβάλλον ε, λόγω του ότι ο περιβαλλοντικό οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου παραμελεί τα καθήκοντά του. Και οικετεύουμε εσά να αναλάβετε δράση, να τιμήσετε τη σύμβαση Άρου, να υπερασπίσετε του πολίτε και να προστατεύετε το περιβάλλον, ε, οδηγώντα τι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου στο δικαστήριο. Σα ευχαριστώ. Πολύ. Η κυρία Γκρός από το από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την τελευταία ενημέρωση του Ιουνίου πήραμε και άλλες πληροφορίες από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς είχαμε ζητήσει να μας δοθούν πληροφορίες για τον υδάτινο ορίζοντα, για το... Ε, ε νερό στο έδαφος τέλος μα, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μα είπαν ότι ήταν μολυσμένο το ε, νερό κάτω από τη χωματερή ε, επιβλήθηκε πρόστιμο 105.000 στερλινών συν ε, δαπάνες ε, καταδικάστηκε λοιπόν ο, ο διαχειριστής της χωματερής αν θέλετε επίσης ε, υπήρχε μια άλλη κατηγγελία ότι ότι ε, χρησιμοποιείται το νερό κάτω από τη χωματερή ε, βεβαίως η ποιότητα του νερού είναι πολύ μεγάλη ε, εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι ε, αφαιρείται το νερό ε, σταδιακά αυτό θα συνεχιστεί και ο δείκτης είναι η περιεκτικότητα σε αμμονία το ο οποίο ελέγχεται. Θα πάρει αρκετό χρόνο για να κατέβει σε νορμάλ επίπεδα η αμμονία. Από εκεί και πέρα θα, για μια άλλη τοποθεσία πιο πέρα θα έχουμε αποτελέσματα σε δύο-τέσσερις εβδομάδες ωστόσο μας λένε ότι παρακάτω στη ροή των υδάτων ε, τα κριτήρια για πόσιμο είδωρ τηρούνται. Άρα δεν έχει επηρεαστεί το νερό. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να ε, ε, επιτρέψουμε τη συνέχιση της λειτουργίας, τη, ε, η απεφασίστη ότι μπορεί να λειτουργήσει η κομματερή για άλλα πέντε χρόνια αλλά μόνο με αναρτή αδρανή απόβλητα και μόνο με απόβλητα νοικοκυριών και όχι βιομηχανικά. Αυτό είναι καλό. Βεβαίως το θέμα έχει πάει και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στην ε, πολεοδομία και βεβαίως και αναμένονται από αποτελέσματα. Εκεί εμπλέκεται βέβαια και μία πλαγιά λόφου που είχε ορυχία. To ask something, if not, it, uh, I'm just shocked that it's more than 10 years that this situation is keeping on. And... Ε, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω η κατάσταση συνεχίζεται. Ο κύριος Βουτσινάρο. Υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά εδώ. Να πούμε πρώτα πρώτα ότι πρόκειται για συγκεκριμένη παραβίαση της οδηγίας West, της οδηγίας, ε, της οδηγίας για τα πόλτα, της οδηγίας για το νερό. Μολύνονται τα υπόγεια ύδατα, αυτό είναι γεγονός. Αυτό επιβεβαιώθηκε από γεωτρήσεις Εφόσον λοιπόν υπάρχουν σαφείς παραβιάσεις, γιατί μετά από δέκα χρόνια πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο γιατί μετά δέκα χρόνια γιατί η Κομισιόν διατηρεί την ηρεμία της και παρακολουθεί με σταυρωμένα χέρια την παραβίαση όλων αυτών των διατάξεων και τι γίνεται με την αρχή Μολύνων πληρώνει διότι εδώ πρόκειται για σαφή υπόθεση, περίπτωση όπου ο Μολύνων πληρώνει για και όχι μόνο για την παραβίαση αυτή καθεαυτή αλλά και για τις παράπλευρες ζημίες για να καθαριστεί η περιοχή κάποια στιγμή. Η κυρία Γκρόσα. Η Κομισιόν εξέτασε την τοποθεσία αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλά ε, δεν προσφύγαμε γιατί διότι για να προσφύγουμε στο δικαστήριο χρειαζόμαστε αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ε, ε, τα παράπονα ήταν ότι η χωματερία αυτή βρίσκεται σε λάθος μέρος. Όντως ε, το να είναι μέσα στη μέση μιας κατοικούμενης περιοχής είναι λάθος. Αλλά από εκεί και πέρα ή είδαμε ότι η σχέση του ε, τοπικού πληθυσμού και των ε, αρχών και των εργολάβων ήταν πολύ κακές ζηκάναμε έρευνες μελετήσαμε τα υπόγεια ύδατα ζητήσαμε από το ε, Geological Survey να κάνει μια έρευνα έγινε αυτό αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο κακά και από εκεί και πέρα έκλεισε η τοποθεσία ε, Βεβαίω οι εθνικέ αρχές προσέφηκαν στο δικαστήριο ε, η οποία επίση καθυστέρησε αλλά ε, στέφθη από επιτυχία γιατί ο διαχειριστή αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμα δεν λέω ότι η κατάσταση είναι τέλεια αλλά δεν μπορούμε ε, δεν μπορεί η Κομισιόν να βασίζεται σε υποθέσεις ή σε ε, καταγγελίες χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εθνικές αρχές προ, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα οι δικές μας οι διαδικασίες δεν είναι για να τιμωρήσουμε να κυρώσουμε, να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κανένα εκείνο που θέλουμε είναι συμμόρφωση και στη τελευταία ανάλυση ποια δεν είναι προς τη αξία αν προσέφευγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικαστήριο Πρόεδρος δεν μπορώ να απαντήσω το ερώτημα, λέει η πρόεδρος. Βεβαίως η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Θέλετε να πείτε κάτι τι. Thank you very much. Να σας ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω κάτι ότι πραγματικά έχω απογοητευτεί τα μάλα τρεις φορές έχουμε έρθει εδώ και τώρα μας λέτε ανοησίες. Όποιος ε, δηλαδή μιλάει εκ μέρους της Κομισιόν μας λέει όλες αυτές τις ανοησίες ε, γιατί πιστεύετε τα ψέματα που σας λένε οι αρχές του ΕΒ για 13 χρόνια. Εμείς ε, δώσαμε το, πάρα πολλές αποδείξεις, 17 τόμους ε, για το τι ε, υφιστάμεθα και πραγματικά είδαμε ότι ρίχνονταν ε, εκεί τα απόβλητα σε ασταθές έδαφος χωρίς να υπάρχει ένα καλό σύστημα στεγανοποίησης και επίσης κλείσανε και το σταθμό άντλησης υδάτων το Μάιο του 2011 γιατί ήταν εντελώς μολυσμένος γιατί σε αυτή τη χαματορή ρίχνουν τα πάντα χημικά απόβλητα ε, λίματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Επίσης, Μα είπαν ότι δεν ρίχνονται εκεί πλέον λίματα από τα νοικοκυριά. Όχι, εγώ μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι ρίχνονται εκεί και είναι και, και καλυμμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διάβασε καν την έκθεση BTS ε, που ήταν αρκετά περιορισμένη και εκεί ε, σχολίαζε ότι υπήρχε περιορισμό και θα μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις ε, που τίθεταν εκεί. Και σε ό,τι αφορά τον, τη συνέχιση ε, της λειτουργίας, ζήτησε άδεια για να συνεχίσει να λειτουργεί χωματερίο φορέας εκμετάλλευσης για 17 ακόμη χρόνια, χωρίς να έχει καμία σχετική άδεια σχεδιασμού. Πραγματικά όλα αυτά είναι σοκαριστικά και οι τοπικές αρχές εν τω μεταξύ έδωσαν ε, άδεια στο φορέα εκμετάλλευσης για να ανατινάξει ένα μεγάλο μέρος της πλαγιάς και αυτό θα οδηγήσει στο να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη τρύπα και αυτό γίνεται στη μέση της πόλης ενώ ο προηγούμενος φορέας εκμετάλλευσης ε, του Λατομείου έκανε ανατινάξεις τότε υπήρχαν ζημίες και πραγματικά η περιβολοντική αρχή δεν ασχολήθηκε καθόλου και μπορώ να σας πω γιατί δεν είμαστε πλούσια περιοχή, είμαστε κανονικοί άνθρωποι, έτσι λοιπόν δεν μετράμε. Και ήρθαμε εδώ ως Ευρωπαίοι πολίτες και σας εμπιστευτήκαμε να μας ε, προστατεύσετε, γιατί δεν το έκαναν οι τοπικές μας αρχές, γιατί για κάποιο λόγο ή για, άλλους, για διάφορους λόγους κάποιοι ε, αξιωματούχοι, κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έκαναν τίποτα να προστατεύσουν, ε, προτιμούν να εξυπηρετούν την πλούσια εταιρεία εμείς ε, ήρθαμε σε εσά, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν ψέματα στην Ευρώπη και έτσι λοιπόν η Ευρώπη αποφάσισε να μην κάνει τίποτα και μάλιστα στη συνέχεια μας έκρυψαν και τα ψέματά τους και εμείς όταν μάθαμε ότι είχαν υποθεί ψέματα τα αποδείξαμε ότι ήταν ψέματα και απευθύναμε μια έκκληση σε εσά, περιμέναμε για 10 χρόνια εσείς να μας βοηθήσετε. Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να αναλάβετε δράση εσείς, γιατί οι δικές μας αρχέ δεν θα κάνουν τίποτα. Υπήρξε μία δίωξη για πέντε κατηγορίες ε, και υπόθηκε ότι η ρήπανση ήρθε από αυτή την διέξοδο υπόγειων ξεκαφημάτων. Βέβαια δεν προήρθε από αυτό. Ε, δεν υπήρχε κανονική στεγανοποίηση ε, της χωματερή. Υπήρχε υποχώρηση των βράχων, γιατί υπήρχε εξόρυξη ε, κάτω από τους βράχους και όταν σταμάτησε να λειτουργεί το ορυχείο μετακινήθηκαν τα βράχια και ουσιαστικά οποιαδήποτε ε, σύστημα πλαστικών μεμβρανών έρχεται εκεί καταραίει. Εγώ πόσο περισσότερο έντονα να σα το παρουσιάσω αυτό. Ήρθαμε εδώ να σα ζητήσουμε βοήθεια, όχι για να μα πει αυτή η ότι πιστεύει ότι τις λένε οι Βρετανικέ αρχέ. Μόνο ψέματα λένε. Σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε την τοποθεσία αυτή το συντομότερο και απευθύνουμε έκκληση στην Κομισιόν να δει το θέμα διαφορετικά. Και σίγουρα θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Ελπίζουμε ότι θα επιληθεί το ζήτημα κατά τη διάρκεια αυτής της συζητίας. Γιατί, ναι, ε, αγωνίσαστε 10 χρόνια και δυστυχώς τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα. Σας ευχαριστώ. Petition number 19. Birds, protection of birds. Πάμε στο σημείο 19 της ε, παραβίασης της προστασίας ε, των θυνών. Όχι, 18 λέει η Πρόεδρος. Έχει να κάνει με την Κύπρο. Ο κύριος Βουτιλιάνο από την Ιταλία. Ο κύριος Ζουτιλιάνο δεν είναι παρόν. Ε, πριν μία ώρα μίλησα μαζί του, μπορώ εγώ να πάρω το λόγο για αυτό το σημείο. Μάλιστα, παρακαλώ. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά στην Κύπρο για την ε, οδηγία προστασίας των άγριων πτηνών ε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Πέρσι το Μάιο εγώ πήγα στην Κύπρο ε, σε ένα σε εκδήλωση κατά της λαθροθυρίας που οργανώθηκε από μια οργάνωση που παρακολουθεί το φαινόμενο αυτό. Παρ' όλα αυτά η ε, σήμερα παρά το ότι η οδηγία απαγορεύει να χρησιμοποιούνται κάποιες ουσίες, ε, σήμερα εξακολουθούν ε, να χρησιμοποιούνται βέργες με κόλλα επάνω ε, για την αχμαλωσία αυτών των πουλιών και χιλιάδες πουλιά αχμαλωτίζονται κάθε χρόνο. Εγώ μίλησα με τον κύριο Τηλιάνο, ο οποίος είναι μέλος αυτής της Ένωσης που έχει έδρα στη Γερμανία, αλλά δραστηριοποιείται και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν εννέα άτομα η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή ε, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές παραβιάσεις ακόμη και αν έχει βελτιωθεί η επαγρύμνηση των τοπικών αρχών ε, σε ό,τι αφορά την περίοδο της Άνοιξης. Υπάρχουν ε, δύο προβλήματα. Η λαθροθυρία την Άνοιξη όπου μεταφέρεται ότι 300.000 πουλιά εκμαλωτίζονται παράνομα και έχουμε και 2 εκατομμύρια πουλιά που εκμαλωτίζονται παράνομα το φθινόπωρο. Υπάρχουν μάλλον αυτή η λαθροθυρία συμβαίνει σε πάρα πολλές τοποθεσίες, ε, κυρίως ε, στο νότιο τμήμα του νησιού, στο κυπριακό τμήμα, στο ελληνοκυπριακό τμήμα. Ε, δυστυχώς δεν αρκούν οι προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου. Επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη ζώνη που ελέγχει το Ενωμένο Βασίλειο. Σε αυτή τη ζώνη ε, έχουμε ε, ουσιαστικά μη δυνατότητα της κυπριακής αστυνομίας να μπει στη ζώνη αυτή και η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε καν ε, πηγαίνει να ελέγξει. Έτσι λοιπόν έχει γίνει ε, μια ζώνη ελεύθερη για τους λαθροθύρες. Ε, και εγώ είδα ότι στα κείμενα της Κομισιόν αναφέρεται ότι υπάρχει δραστηριότητα επαναπτύσσεται από τις δύο αρχές, αλλά σας διαβεβαιώ οι εθελοντές μου είπαν ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Υπάρχει πραγματική ανοιχτή ανοχή της λαθροθυρίας σε αυτή την περιοχή. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ενήμερες ε, γιατί από ό,τι φαίνεται η Wildlife Crime Unit ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, πρόσφατα εκπώνησε μία έκθεση όπου εντοπίζεται το πρόβλημα αυτό. Σε ό,τι αφορά στο έγγραφο εργασίας της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται ότι στην Κύπρο υπάρχει υπάρχει ε, ουσιαστικά μια νομοθεσία που επιβάλλει κυρώσεις ε, του ύψους, πρόστιμα του ύψους 17.000 ευρώ στους λαθροθύρες. Ε, εγώ στην Ιταλία ήμουν ε, εθελοντής, ε, ε, συνεργάστηκα με τι τοπικέ αρχές ε, κατά, για την καταπολέμηση της ελευθερωτηρίας. Ε, ήμουν εθελοντής φύλακα. και μπορώ να σας πω αν οι αρχές της Κύπρου ακόμη και αν λένε ότι θέλουν να καταπολεμήσουν την ελευθερωτηρία τελικά το αντίθετο συμβαίνει. Μιλώντας ψυχολογικά οι ελεγκτικές αρχές ε, μπροστά σε ένα τέτοιο δίκημα για το οποίο προβλέπεται πρόστιμο της τάξης των 17.000 ευρώ. Ε, τι να σας πω, δεν είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Θα ήταν ε, καλύτερο ε, να υπάρχει ένα πρόστιμο 2-3.000 ευρώ γιατί να επιβάλλει κανείς ένα πρόστιμο 17.000 ευρώ σε έναν ε, πολίτη θα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Έτσι λοιπόν αυτή η κύρωση ε, οδηγεί τις αρχές να μην επιβάλλουν τελικά, το ύψος αυτής της κύρωσης οδηγεί τις αρχές να μην επιβάλλουν τελικά αυτό το πρόστιμο αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να παρακολουθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να ξεκινήσει και διαδικασία επί Γιατί αν το κράτο μέλο δεν ε, εγγυάται του απαραίτητου ελέγχου και κυρίω ε, το φθινόπωρο το βλέπουμε αυτό, Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία επί και να μην ξεχνάμε ότι η Δία ε, των Πτηνών είναι μία από τις ε, πρώτες ε, οδηγίες για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μεριά της Επιτροπής παρακαλώ ο κύριος Good morning. Thank you, Mr. Um, I would be... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καλημέρα θα είμαι σύντομος γιατί σχετίζεται με το γενικότερο θέμα της λαθροφρίας σε πολλές άλλες χώρες. Ε, προς το παρόν θα ήθελα... No, I will be brief on issue. Are... I can be briefly. Okay. Uh, I can briefly inform you about this issue. Ειδικά για αυτό το θέμα της Κύπρου θα πω πολύ λίγα πράγματα και μετά θα αναφερθώ στο γενικότερο θέμα στην Ευρώπη. Λοιπόν, για την Κύπρο πρώτα-πρώτα το θέμα είναι πολύ γνωστό. Πρόκειται για παράνομες πρακτικές ε, βάσει του κοινοτικού δικαίου αλλά και βάσει του κυπριακού δικαίου. Ε, μακρόχρονη ιστορία με πολυδιάστατη οικονομική, κοινοτική κοινωνική, πολιτική κλπ. Και η Κομισιόν παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση ακόμη από την εποχή πριν να ενταχθεί και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέρα για να βελτιωθεί η σύμμορφη εφαρμογή ε, για να μην χρησιμοποιούνται πια οι βέργες και τα δίχτυα και ε, Υπάρχουν βεβαίως κάποια συγκεκριμένα βήματα που ήδη έχουν γίνει όχι μόνο από τις κυπριακές αρχές αλλά και από τις αρχές της βρετανικές, της βάσης όπου βεβαίως δεν ισχύει το κοινοτικό κεκτημένο αλλά ε, ε, ε, εφαρμόζεται και εκεί υπάρχει ανάγκη σωστής εφαρμογής παντού με άλλα λόγια κάτι τι έχει γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση έγιναν έλεγχοι επιτόπου έγινε κατάσχεση όλων αυτών των παράνομων εργαλείων ε, υπάρχει και καινούργια νομοθεσία που επιβάλλει και πρόστιμα υπάρχει καλύτερο συντονισμό των διαφόρων αρχών και με την αστυνομία και με τις αρχές που ασχολούνται με το κυνήγι και με τις αρχές στο βρετανικό τομέα και βεβαίως υπάρχουν και πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί προστασίας περιβάλλοντος που είναι πολύ ενεργοί, πολύ δραστήριοι. Υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα στην, κατά τη διάρκεια της αρινής μεταναστευτικής περίοδου των πτυνών αυτών είδαμε να βελτιώνονται τα πράγματα. Ωστόσο, όπως είπε μόλις ελέγχθη, το φθινόπωρο είναι κακή η κατάσταση, το φθινόπωρο είναι κακή η κατάσταση, συνεχίζει να είναι κακή. Και εκείνο που θέλω να πρόκειται να κάνουμε είναι να ξαναέρθουμε σε επαφή με τις Κυπριακές και τις Βρετανικές αρχές για να κουβεντιάσουμε αν μπορούν να πάρθουν επιπλέον μέτρα για να υπάρξει πραγματική βελτίωση και το φθινόπωρο. Και βεβαίως δεν αποκλείεται προσφυγή επί στο δικαστήριο ε, αν και εφόσον δούμε ότι οι αρχές δεν ενδιαφέρονται αλλά όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και σε άλλα μέρη της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντιμετωπίσει με ένα ολιστικό τρόπο το θέμα. Επόμενη αναφορά Μάλτα, Κύπρος και άλλες χώρες. Κύριος Ρώτη, παρακαλώ. Goedemiddag ondertussen, dames en heren. Voor eerst wil ik u in naam van de Belgische... Θα ήθελα εκ μέρου τη Ένωσή μα να σα ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση σχετικά με την αναφορά μας και την σφαγή πτηνών στη Μάλτα. Υπάρχουν μεταναστευτικά πτηνά που διασχίζουν εκτάσεις, πετούν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα για να μπορέσουν να διαχυμάσουν κινδυνεύουν να χαθούν, κινδυνεύουν το κρύο, κινδυνεύουν από τη έλλειψη τροφής και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εάν δεν τα καταφέρουν θα πεθάνουν στο δρόμο. Πολλά τέτοια πτηνά κινδυνεύουν επίσης από αρπακτικά ή άλλα πτηνά. Οι φυσικές απώλειες λοιπόν είναι σημαντικές αλλά λελογισμένες. Αρκετά δηλαδή πτηνά επιβιώνουν για να διονυστεί το είδος. Στην Ευρώπη τα πτηνά αυτά δυστυχώς κινδυνεύουν και από τον άνθρωπο. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Πολλά από αυτά όπως προείπα είναι μεταναστευτικά. Οι άνθρωποι τα κυνηγούν κατά μήκος της Μεσογείου. Δυστυχώς οι σφαγευτοί είναι ομαδική. Στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στη Μάλτα, στην Κύπρο κάθε χρόνο εκατομμύρια πουλιών βρίσκουν τον θάνατο εξαιτία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μόνο στη Μάλτα κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστευτικά πτηνά παγιδεύονται, σκοτώνονται παρά το γεγονό ότι είναι προστατευόμενα. Σε διάφορα κρατημέλη έχουμε προγράμματα για την προστασία ακριβώ αυτών των φυτών των πτηνών, με συγχωρείτε. Η Μάλτα είναι ενδιάμεσος σταθμό του σπίν για τα πτηνά αυτά, τα φθινόπωρο. Αντί να βρουν εκεί λοιπόν καταφύγιο στην Μάλτα, τα πτηνά αυτά αντιμετωπίζουν μια ομαδική σφαγή, ενώ ανεβαίνουν από τις νοτιότερες περιοχές προς τα βόρεια. Χιλιάδες κυνηγοί λοιπόν τους επιτίθενται, κατά μήκο των αποκριμνών ακτών της Μάλτας. Οι ακτές αυτές γεμίζουν ε, παγίδες, ξόβεργες, δίκτυα και σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 3 εκατομμύρια πτηνά το φθινόπωρο παγιδεύονται στην περιοχή και τίθενται σε κλουβιά. Αποτελεί πλέον παράδοση στην Μάλτα. Τα πουλιά αυτά στη συνέχεια πολλούνται. Το 2012 η BirdLife Malta, η οργάνωση BirdLife Malta, περιμάζεψε 101 τραυματισμένα ή νεκρά πτηνά. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, ο μεγαλύτερος τα τελευταία χρόνια, που δείχνει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Φυσικά τα τραυματισμένα πτηνά αποτελούν ένα πολύ μικρό κλάσμα αυτών που συλλαμβάνονται ή θανατώνονται. Η BirdLife Malta ε, έχει δημιουργήσει διάφορες επιθεωρήσεις και διαπίστωσε ότι πολλά πτηνά εχμαλωτίζονται παρανόμως. Έχουμε βεβαίως και το κυνήγι με πυροβολά όπλα, πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα να λάβει κανείς υπόψη του ότι υπήρχε και σύμφωνα μεταξύ του Εργατικού Κόμματος και των κυνηγών πριν από τις εκλογές. Αυτό είχε παρουσιαστεί ως μια απόπειρα να αποστρεφθούν οι καλλιέργειες από τα πτηνά. Στην Μάλτα υπάρχει βεβαίως άδεια θύρας. Η χορήγηση όμως της ε, άδεια αυτή έχει γίνει πολύ πιο εύκολη. 9.500 κυνηγοί ενεγράφησαν πριν από την Άνοιξη φέτος ενώ πέρσι ο αριθμός αυτός ήταν 6.000. Για να ελεγχθούν αυτοί οι κυνηγοί θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 66 αστυνομικού. Η θηροφυλακή δυστυχώ έχει μόνο 16 έλεγκτε. Είναι προφανέ ότι δεν είναι δυνατό ο αποτελεσματικό έλεγχο εν προκειμένου. Όπω έλεγα, διευκολύνεται η διαδικασία απόκτηση κυνηγητικού όπλου, οι έλεγχοι είναι λιγότεροι και λιγότερο αποτελεσματική, όλα συντείνουν στο συμπέρασμα ότι η Μάλτα δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει το παράνομο αυτό κυνήγι. Και το οποίο και εξηγεί με τη σειρά του το καταστροφικό αποτέλεσμα που έχουμε και θα έχουμε το 2013. Δεν έχουμε καμία ένδειξη σύμφωνα με την οποία οι αρχές ε, προτίθενται να κάνουν κάτι. Όλο μάλλον να πάρουν ριζοσπαστικά μέτρα ελέγχου. Διερωτώ στην περίπτωση της αστοχίας της κυβέρνησης να λάβει μέτρα, εάν η Κομισιόν λοιπόν σκοπεύει να ζητήσει από τις αρχές της Μάλτας να λάβουν τα επιβαλλόμενα μέτρα. Δεν θα έπρεπε να παρέμβει η Κομισιόν για να προλάβει την εξαφάνιση εκατοντάδων χιλιάδων πουλιών διαφορών Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Ευχαριστώ. Καταρχήν, να επενθυμίσω ότι σε σχέση με τη Μάλτα υπήρξε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2009 που άφησε ανοιχτή τη δυνατότητα να υπάρχει μια παρέκκληση για δύο, η θηθήρα δύο ειδών. Αν λάβουμε υπόψη τις συνθήκες ε, στη Μάλτα, προβλέπεται και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ε, αρινή περίοδο στην Εθνική Νομοθεσία. Η Εθνική Νομοθεσία δηλώνει ότι ε, είναι περιορισμένος ο αριθμός ε, των πτηνών που ε, θυρεύονται το φθινόπωρο και επίση επιτρέπονται να θυρεύονται περισσότερα την άνοιξη. Επίση, περιλαμβάνονται κάποιε ποσοστώσει και περιορισμοί σε σχέση με τον τρόπο και τον χρόνο σε ό,τι αφορά την ε, έναρξη της φετινής ερνής περίοδου, ενημέρωση μάλιστα την Κομισιόν ε, μέσω του αρμοδί, της αρμόδιας υπηρεσίας ε, και επίσης θεωρήθηκε ότι πληρούνταν οι προποθέσει για να δοθεί παρέκκληση και φέτο στη Μάλτα. Η Κομισιόν ε, σημείωσε την απόφαση των αρχών της Μάλτας ε, ε, βέβαια θέλουμε να υπάρχει κατάλληλη παρακολούθηση επιτόπου έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζεται σωστά η παρέκκληση. Η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητες να παρέμβει ε, για να αναστείλει ή να σταματήσει την ε, θύρα κατά τη διάρκεια της περίοδου, γιατί αυτό η απόφαση λαμβάνεται από την κυβέρνηση. Θέλω πάντως ε, να υπενθυμίσω ότι τα κράτη-μέλη στέλνουν εκθέσεις στην Κομισιόν και για τη Μάλτα επίσης πρέπει να υποβληθεί αυτή η έκθεση για να δείξουμε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την παρέκκληση και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστά τα όρια της παρέκκλησης Επίσης, μπορούν ε, οι εκθέσεις αυτές ε, να σταλούν ε, και από άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις και πρέπει φυσικά να αποδεικνύεται ότι γίνεται σεβαστή η οδηγία για την προστασία των άγριων πτηνών. Επίσης, τα εθνικά όργανα είναι αρμόδια για να καταπολεμήσουν παράνομες πρακτικές όπως ε, η λαθροθυρία. Τα τελευταία χρόνια η Μάλτα άρχισε να παίρνει κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσει το θέμα, όπως το χάρη κυρώσεις ε, έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και έχουν σημειωθεί και κάποιες ε, δικαστικές διώξεις. Παρόλα αυτά, η παράνομη θανάτωση ε, των πτηνών στη Μάλτα την άνοιξη του φθινόπωρο προκαλεί ανησυχία και η Κομισιόν περιμένει η κυβέρνηση της Μαλτάς να συνεχίσει τις προσπάθειες για να αποτρέψει τις πρακτικές και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας θα οδηγήσει σε προσφυγή στα δικαστήρια. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παράνομες πρακτικές ε, που πλήττουν ε, τα πτηνά, όχι μόνο η παράνομη θανάτωση, αλλά και η παράνομη παγίδευση και η δηλητηρία, συλλαμβάνουν χώρα όχι μόνο στη Μάλτα αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Επομένως, η Κομισιόν συμφώνησε στη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και τα διαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, να καλύψει μίσο, όπως η, η παρακολούθηση παράνομων δραστηριοτήτων, ανταλλαγή πληροφοριών ε, και ε, βελτίωση της πρόληψης. Ε, πρέπει να εφαρμοστούν ε, οι εντοπισμένε δράσει από τα κράτη-μέλη τη stakeholders ή την Κομισιόν. Επίση, η Κομισιόν ξεκίνησε μια συνεργασία με το λεγόμενο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και φυσικά επικεντρωνόμαστε στο θέμα της παράνομης θανάτωσης και παγίδευσης και αχμαλωσίας ε, των πουλιών και θα γίνει μια συνεδρίαση στη Μάλτα τον Οκτώβριο Κομισιόν. Δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μάλτα και θα συνεχίσουμε το διάλογο με τις αρχές της Μάλτας προκειμένου να προσδιορίσουμε περαιτέρω βήματα που ίσως πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των άγριων πτηνών. Ευχαριστώ. το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά στη Μάλτα, επίσης είναι γνωστή αυτή η κατάσταση παρανομίας που διαρκεί χρόνια. Έχουμε παραβίαση της οδηγίας ε, περί προστασίας των πτηνών και από την πλευρά της μαλτιστικής κυβέρνησης ε, υπάρχει ουσιαστικά εντελώς ε, έλλειψη σεβασμού και αυτή την οδηγία. Εγώ επί τόπου ε, συμμετείχα σε ένα καταβλισμό λαθροθυρίας το Σεπτέμβριο του 2012 και είδα τι συμβαίνει. συμμετείχα με την Bird Life της Μάλτας και με την Επιτροπή κατά τους θανάτωσης των πτηνών. Οι κυνηγοί έχουν αυξήσει τη λαθροφυρία και τώρα στη Μάλτα που είναι με της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε ε, σε περίοδο άνοιξης ε, και ξέρετε ε, τα πουλιά ε, κυνηγούνται στη Μάλτα ενώ βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής και συγκεκριμένα κυνηγούνται τα τριγώνια και τα ορτίκια. Τι έκανε η Μάλτα ε, φέτος με δύο ε, νόμους για να επιτρέψει το κυνήγι στην άνοιξη από τις 10 ως τις 30 Απριλίου και αποφάσισε να εφαρμόσει τι παρεκκλήσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έχουν καταργοποιηθεί 16.000 ε, κατηγορίε πτυνών. Ε, ε, υπάρχουν 9.000 κυνηγοί στη Μάλτα και επέτρεψαν 20 μέρε θύρα. Και επειδή, όπως σας είπα και στη χώρα μου, έχω επιδοθεί σε δραστηριότητες φύλαξης κατά της λαθροθυρίας, ήδη ε, έχουν φτάσει στη Μάλτα στο όριο, όχι την πρώτη μέρα, αλλά τις πρώτες ώρες της θύρας. Δεν χρειάζεται η Κομισιόν λοιπόν καμία έκθεση, δεν χρειάζεται τίποτα, γιατί ήδη στην νομοθεσία υπάρχει υπάρχει ε, τελικά μια κοροϊδία σε Ένωση τη Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Τελικά μα κοροϊδεύουν γιατί αυτά τα νούμερα, σε αυτά τα νούμερα φτάσανε σε αυτά τα όρια μέσα σε δύο-τρει ώρε. Έτσι λοιπόν ε, τελικά η Κομισιόν πρέπει να παρέμβει για να κάνει αυτό το κράτο μέλο να καταλάβει ότι η οδηγία των πτηνών είναι μία από τι πιο παλιέ οδηγίε που θα πρέπει και αυτοί να τη σεβαστούν δεν πρέπει πια να μας κοροϊδεύουν. Η προεκλογική τους εκστρατεία ε, συμπεριλάμβανε και τέτοιες υποσχέσεις ε, και τελικά απελευθέρωσαν ε, εντελώς ε, την περσινή παρέκκληση. Στο άρθρο 9 έχουμε τις ε, μικρές ποσότητες. Δεν το έχουν σεβαστεί, δεν υπάρχουν έλεγχοι, γιατί δεν υπάρχουν φυσικά οι δυνάμεις από την αστυνομία για να ελέγξουν 9.000 κυνηγού. Και αυτό όλο τι σημαίνει, όχι μόνο ότι δολοφονούν αυτά τα δύο είδη, αλλά απόλυτη λαθροθυρία επί όλων των ειδών που είδατε στις διαφάνειες. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυνηγούν ό,τι κινείται. Έτσι λοιπόν, ε, σας επαναλαμβάνω, οι αρχές ε, δεν θέλουν καν να κάνουν ελέγχους, το έχουν, ελέγχους, το έχουν πει ξεκάθαρα. Όμως ο νόμος πρέπει να είναι ο ίδιος ε, για όλα τα κράτη-μέλη και για τη Μάλτα. Και η μόνη γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι είναι οι κυρώσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μια διαδικασία επί παραβάση. Ας υπάρχει και άλλη μια καταδίκη με κυρώσεις η πρώτη απόφαση που υπενθυμίσατε, που επέτρεπε αυτή την παρέκκληση, την επέτρεπε δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας, αν γινόταν σεβασμό το άρθρο 9. Όμως ε, εδώ έχει καταστρατηγηθεί εντελώς. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν 7 αναφορές ε, για αυτό το θέμα. Όλοι οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται. Εγώ έκανα μια ερώτηση στην Κομισιόν πριν λίγες ημέρες για να ζητήσω παρέμβαση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έλαβα πάρα πολλά email και τηλεφωνήματα από πολίτες από όλη την Ευρώπη, γιατί πραγματικά έχουν σοκαριστεί. Υπάρχουν 7 ε, αναφορές για αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να χάνουμε άλλο χρόνο και ε, πρέπει να είμαστε ουσιαστικά να αντιδράσουμε, να μην επιτρέψουμε η κυβέρνηση της Μάλτας να μας κοροϊδεύει. Η Επιτροπή ε, μας θα φροντίσει να πιέσει λίγο την Επιτροπή, την Κομισιόν προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία την οποία προτείνεται. Τέλος πάντων θα το συζητήσουμε και με τους συντονιστές. Την κρατούμε ανοιχτή, δεν το συζητάμε, άλλωστε αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Ε, προχωρούμε... Α, yes, Mr. Sorry. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά εκπρόσωπα της Κομισιόν, η Ρουμανία, η χώρα μου, έχει την ε, μεγαλύτερη περιοχή βιοπικιλότητας στην Ευρώπη, το Δέλτα του Δούναβη. Και με αυτό που αναφέρετε πριν, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, αν εφαρμοζόταν αυτή η πρακτική, θα είχε καταστραφεί εντελώ το Δέλτα του Γιατί δεν έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά η Κομισιόν, δηλαδή να υπάρχει επαρκής προστασία μεν για το δέλτα του Δούναβη για να αποφεύγονται οποιασδήποτε ζημίες ε, κατά της βιοποικιλότητας του Δούναβη ενώ ταυτόχρονα ε, δέχεστε τη θανάτωση των πτηνών γιατί όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και στη Μάλτα είναι σφαγή των πτηνών. Τι προσπαθείτε να μας πείτε. Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν όρια, προσπαθούν να ε, σταματήσουν, ε, να αποτρέψουν τη θανάτωση. Ωραία όλα αυτά τα λόγια, αλλά εντελώς μη ρεαλιστικά. Και να σας πω κάτι ακόμα. Υπήρξε δυνατότητα να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Καταρχήν υπήρξε ε, έρευνα από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή κοντά στο ΔΕΛΤΑ του Δούνεβη για τον πολύ απλό λόγο και εγώ υποστήριξα τη δράση της Κομισιόν, έγινε μια τέτοια απόπειρα, γιατί ε, εκεί ε, θεώρησαν ότι αιωλικά πάρκα που επρόκειτο να εγκατασταθούν εκεί, ότι αυτά θα ενοχλούσαν την πορεία των μεταναστευτικών πουλιών όταν από τον Νότο πήγαιναν στο Βορρά. Έτσι λοιπόν, εμείς ε, στη Ρουμανία πρέπει να ξοδέψουμε και μερικά από τα ευρωπαϊκά χρήματα για να προστατεύσουμε τα μεταναστευτικά πτηνά, μεν, ενώ εσείς ε, δεν δέχετε και μάλιστα έχετε και συνένοχη θα έλεγα να γίνεται τέτοια σφαγή πτηνών, θανάτωση πτηνών στην Κύπρο και στη Μάλτα. Πείτε μου κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν, πού είναι η συμμεταχείριση εδώ. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατό σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Αφρική, όχι σε περιοχές όπου έχουμε σαφάρι, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτρέπεται μια τέτοια μεταχείριση. Οι δύο χώρες που προαναφέρθησαν είναι κρατημέλη. Ξέρω πολύ καλά ότι με το σημερινό τεχνικό εξοπλισμό μπορούμε να δούμε πεταλούδες, έντομα. Συγγνώμη, αλλά είμαι εξοργισμένος, κυρία Πρόεδρε. Γιατί είναι απαράδεκτο να μην βλέπουμε πότε θανατώνονται τα πουλιά και να μας λέει η Κομισιόν. Μα υπάρχουν ειδικέ συμφωνίες, υπάρχουν διατάξεις μεταβατικές κτλ. Όλα αυτά είναι λόγια. Η Κομισιόν θα έπρεπε να εφαρμόζει διάμετρα και σταθμά όπως αυτά ισχύουν στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Δούναβη. Διαφορετικά για τη Ρουμανία να ξοδεύει περισσότερα χρήματα ή να έχει τόσο υψηλό αριθμό πτηνών μεν και να σκοτώνονται άνθρωποι στη Ρουμανία. Πείτε μου, πού είναι η συμμεταχείριση. Διαφορετικά να κάνουν και τα άλλα κρατημέλη ειδικέ διευθετήσεις με την Κομισιόν και να επιτρέπεται αυτή η θανάτωση. Είναι εντελώ απαράδεκτη λοιπόν αυτή η κατάσταση. Uh, let's go to the next... Uh, Ας συνεχίσουμε. Ας περάσουμε στο επόμενο ή όχι. Χιλκλέν. Όσον αφορά την κράση στη Μάλτα, την Άνοιξη και το φθινόπωρο, που έχουμε λιγότερα ε, πουλιά, οι ε, κυνηγοί βαράνε ότι πετάει όταν δεν υπάρχουν μεταναστευτικά πτηνά. Οι κυνήγοι λοιπόν θα κυνηγήσουν ε, λιβελούλες, πεταλούδες, ό,τι βρουν, εν πάση περιπτώσει. Την άνοιξη οι κυνηγοί ασκούνται στα χελιδόνια. Διάφορα είδη χελιδονιών τα οποία επιστρέφουν από την, τις του Κονγκό ανεβαίνοντας προς την Ευρώπη. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ. Uh, Το κρατάμε λοιπόν ανοιχτό. Κύριε Μποστινάρου, κρατάμε αυτά που είπατε σχετικά με τα ποιοτικά μέτρα και να περάσουμε στην επόμενη Μποστινάρου. Να στείλουμε τις αναφορές και στην Επιτροπή ΕΝΒΙ γιατί Πρέπει να ζητήσουμε μέτρα διόρθωσης αυτή της κατάστασης. Πολύ καλή ιδέα λέει. Πρόεδρος θα το κάνουμε. Ε, ένδικα, ε, να χρησιμοποιηθούν και ένδικα μέσα. Πολιτική μεταφορών της Ιρλανδίας από την... Ε, ο κύριος Κάνιφ. Α, there you are. No, there you are. I wish to thank Madam President and the committee members Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ σήμερα. Ε, η Δυτική Αψίδα συνδέει έξι πόλεις της Ιρλανδίας. Ε, ε, εδώ δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε ε, το σιδηρόδρομο που βρίσκονται στη Δικευσίδα, αλλά ε, εδώ θέλουμε να μιλήσουμε για την έλλειψη διαφάνειας στη χρήση των κονδύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αποφάσεις ε, πολιτικής μεταφορών στην περιοχή BMW. Η Ιρλανδία είναι μία από τις ε, πιο κεντρικές οικονομίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στο Δουβλίνο βρίσκονται όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Τα προγράμματα του 2006 Είδα πάνες οι κυρίες δαπάνες ε, για ε, τις μεταφορές ε, έγιναν στο Δουβλίνο. Όμως τα γεγονότα δεν σταματούν να υπάρχουν επειδή τα αγνοούνται. Αυτό το είπε ο Άλντους Χάξκλεϊ. Και σε απάντηση στην Κομισιόν το ΕΤΠΑΣ έχει εγκρίνει σημαντικές επενδύσεις για τις μεταφορικές υποδομές της Ιρλανδίας και δέσμευσε χρηματοδότηση για κάθε περιοχή, όμως δεν έγινε σεβαστή η κατανομή του ΕΤΠΑ. Αυτή είναι μια σοβαρή παραβίαση που πρέπει να διερευνηθεί και ουσιαστικά τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί για την περιοχή BMW της Ιρλανδίας παρεκτράπησαν για κάποια άλλα project ε, για την πιο πλούσια νότια και ανατολική περιοχή στο πρόγραμμα 2000-2006. Ε, στην περιοχή BMW ε, δεν έχουμε λάβει συγκεκριμένη κατανομή ανατμήμα για το πρόγραμμα 2000-2006. Είναι βέβαιο ότι δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια διαβούλευση σε σχέση ε, με το TNT ε, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ε, μεταφορών ε, από τα οποία έχει αποκλειστεί η όλη περιοχή. Χρειαζόμαστε περισσότερες συνδέσεις με αυτοκινητόδρομους για συνοριακά και σιδηροδρόμους προκειμένου να υπάρξει οικονομική μεγέθυνση. Θέλουμε επίσης περισσότερη διαφάνεια για τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για την περίοδο 2014-2020. Στην Ιρλανδία δεν έχει γίνει καμία ανάλυση κόστους οφέλους για τη δυνατότητα διασυνοριακού έργου ε, στην ε, περιοχή BMW και αυτό ουσιαστικά παραβιάζει τις αρχές διαφάνειας και είναι κατά το κατευθυντήριο γραμμών TNT. Ε, Επίσης, ε, ε, στα προγράμματα όπου υπάρχει χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει καλύτερη εξέταση και αξιολόγηση, γιατί διαφορετικά θα καταπατήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mr. Langley. Yeah, I'm here. Okay, thank you. Um... Ευχαριστώ. Μέλη της Επιτροπής. Είμαι ο Πίτερ κτηνίατρος από αυτήν την περιφέρεια της Ευρώπης. Πιστεύω ότι οι βασικές αρχές της δημοκρατίας, αλληλεγγύης και συνοχής πρέπει να διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που εξασφαλίζουν τις ευκαιρίες στους πολίτες της Ευρώπης ως ε, χειρουργός ε, κτηνίτρος. Υπόκειμε σε κανόνες. Οι κανόνες υπάρχουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να απολαύουν όλοι ίσων ευκαιριών, είναι ζωτική σημασία να υπάρχει δικαιοσύνη και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συναλλάσσονται. Ιδιαίτερα όταν ε, χορηγούν ευρωπαϊκά κονδυλία η οργάνωσή μας, χωρίς να έχει κομματικές ε, προσβάσεις, θεωρεί ότι δεν τη χάνουμε ισοτιμής μεταχείρισης. Χρειαζόμαστε υποδομές στην περιοχή μου για να αντιμετωπίσουμε και κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Χρειαζόμαστε λοιπόν στα βορειοδυτικά την απαραίτητη υποδομή για να ανασταλεί η οικονομική και η κοινωνική αιμορραγία που επηρεάζει οικογένειε και τον τοπικό Το χρειαζόμαστε για τι επόμενε γενναίε. Για να μπορέσουν οι επόμενε γενναίε να συνεχίσουν να συνεχίσουν να επιβιώνουν με συμβασμό. Το δυτικό τόξο είναι ένα έργο το οποίο θα άρει τις ανισότητες που πλήττουν την περιοχή μας και την Βόρεια Ιλανδία γενικότερα. Θα βελτιώσει την κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν και θα φέρει πιο κοντά τις ε, περιοχές της περιφερειάς μας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, η οποία ανακήρυξε αποδεκτή την αναφορά μας. Ευχαριστώ πολύ. Madam President, my name is Paul O'Connor. Κύριε Πρόεδρε, Paul O'Connor. Ζω στα βορειοδυτικά της Ιρλανδίας. Έχω μια μικρή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε μέσα στην ύφεση. Χρειαζόμαστε υποδομές. Έχουμε μορφωμένους εργαζομένους. Το μόνο που μας λείπει είναι επαρκείς υποδομές. Κάτι το οποίο θα ενθαρρύνει νέες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην βορειοδυτική ακτή της Ιρλανδίας. Θέλουμε να δώσουμε τέρμα στις ανισότητες που πλήττουν την περιφερειά μας. Προσωπικά εμείς στην περιοχή βρισκόμαστε σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ακριβώς επειδή δεν είμαστε μέλη των προγραμματών ΤΑΦ 10, των διευρωπαϊκών δηλαδή δικτύων. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Έφυγα από την Ιρλανδία και δούλεψα σαν στέλεχος επιχειρήσεων στην Αμερική και αλλού. Γύρισα όμως πριν από μερικά χρόνια στην Ιρλανδία και ασχολούμαι τώρα με τον τουρισμό στην ε, δυτική ακτή της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τουρισμός, ιδιαίτερα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ιρλανδία. 90% των Ευρωπαίων τουριστών κυκλοφορούν με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Είναι λοιπόν αδύνατον να αγνοήσουμε τις ελλείψεις αυτές που υπάρχουν στη χώρα μου ε, δεν μπορούμε να ε, συνεχίσουμε με αυτό το μειονέκτημα την έλλειψη σωστών δικτύων διότι αυτό μας βάζει σε δυσχερέστερη σχέση και σε σχέση με το τουρισμό, με την ανατολική πλευρά κτλ. Επίσης η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων είναι πολύ σημαντική και αυτό και επηρεάζεται από την έλλειψη δικτύων στην περιοχή μας. Υπάρχουν και άλλα θέματα και κοινωνικά και θέματα ιατρικής περίθελψης ε, και αυτά παρεμποδίζονται με δεν υπάρχουν τα σωστά μέσα μεταφοράς. Το ίδιο και στα... για θέματα παιδείας για τους νέους. Αυτό είναι ένα επιπλέον εμπόδιο για τη σωστή τους εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχουμε ψηλό επίπεδο κατάρτιση, αλλά το να μην ε, ε, έχουν κάποιοι σπουδαστές πρόσβαση εκεί που θέλουν να πάνε γιατί δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς αυτό είναι κακό και για τους σπουδαστέ και για τους νέους και για οποιαδήποτε ηλικία πολίτες είναι αδικαιολόγητη η κατάσταση αυτή. Επίσης υπάρχει αδιαφάνεια στη διαδικασία λήψης απόφασης και εκ μέρους όλων αυτών των πολιτών, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, σα ζητώ να βάλετε την Ιρλανδία, την περιοχή μας, στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ή οφείλουμε κάποιες υπηρεσίε στους πολίτες μας. Και τέλον τελειώνοντας να ευχαριστεί να σας ευχαριστήσω και σας και την Επιτροπή σας που κάνατε παραδεκτή την αναφορά μας σας ευχαριστώ. Λάγκλη. Ο κύριος Λάγκλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν κάμποσα θέματα που θα μπορούσα να σχολιάσω. Μερικά από αυτά προσπαθήσαμε να τα καλύψουμε στην αρχική μας απάντηση προς την αναφορά αυτή. Πρώτα πρώτα το θέμα των διαβουλεύσεων διότι εδώ υπάρχει μια ανακρίβεια στο τι είπαμε στην επίσημη απάντησή μας για την δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πρόγραμμα για υποδομές 2000-2006 και εκείνη την περίοδο έγινε και δεύτερη διαβούλευση διαβούλευση όμως κατά κύριο λόγο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που λειτουργούν το σύστημα κοινωνικών εταίρων της Ιρλανδίας. Δεν ήταν πραγματική δημόσια διαβούλευση αυτή. Αυτά για το 2000-2016. Αλλά για το επόμενο πρόγραμμα, το περιφερειακό, το 2007 μέχρι το 2013, επιβεβαιώνεται στα έγγραφα αυτά καθεαυτά δικτύου προγράμματος ότι έλαβε χώρα δημόσια διαβούλευση και έχω εδώ μπροστά μου και βεβαίως μπορώ να το δώσω και στους αναφέροντες ένα παράδειγμα για τη συμπεριλήψη όλου ή μέρους του δυτικού ο, διαδρόμου ε, στις προτάσεις ε, που έγιναν. Αυτό δεν το δέχτηκαν οι Ιρλανδικές αρχές και αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Θα επανέλθω σε αυτό και θα σας πω γιατί σε μερικά λεπτά. Οι αναφέροντες ε, μίλησαν για την ε, ε, κατανομή, τη λεπτομερή περιγραφή των ε, προγραμμάτων για την περιοχή τους την τελευταία προγραμματική περίοδο βεβαίως αυτή η περίοδος συνεχίζεται και κάνουμε πράγματι λεπτομερή απαρίθμηση και περιγραφή των προγραμμάτων αυτά τα αυτοί οι κατάλογοι μπορούν να σας δοθούν βεβαίως. Άρα γίνεται καταγραφή λεπτομερής. Δεύτερο θέμα. Βεβαίως από το 2008 η Ιρλανδία βρίσκεται σε κρίση, έχει προβλήματα και το 2009 είδαμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε σε ορισμένα σημεία το πρόγραμμα. Μέρος του δυτικού διαδρόμου θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί. Αυτό το παρουσίασε η διαχειριστική αρχή αλλά μετά αποφασίστηκε, φαντάζομαι από το Υπουργείο Μεταφορών, ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί η χρηματοδότηση αυτή. Εκείνο που μας είπαν οι Ιρλανδικές αρχές είναι ότι υπήρχε θέμα κόστους οφέλους εδώ. Δηλαδή ότι άλλο θα ή πριν να χρηματοδοτηθεί κάποιο πρόγραμμα πρέπει να αποδειχθεί η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος και θα πρέπει να καταδειχθεί επίσης ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν ο δυτικός διάδρομος δεν συμπεριελήφθη τα μία από τις πιθανές επενδύσεις κατά την τροποποίηση του προγράμματος. Επίσης υπάρχουν άλλα δύο βασικά σημεία υποδομής, οδικής υποδομής που συμπεριλήφθησαν αυτοκινήτων ένα κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου του αυτοκινητοδρόμου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλο ένα ε, κομμάτι για τα bypasses. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε να δούμε μπορούμε να κάνουμε στα προγράμματά μας και στο 2007 2013 και στο 2014 2020 ε, θα δείτε ότι δεν προβλέπονται μεγάλα κονδύλια για την χρηματοδότηση των μαζικών μέσων συγκοινωνιών μεταφορών στην Ιρλανδία. Δεν προβλέπεται στο μέλλον. Τώρα για τα τέντ, τα δίκτυα αυτά. Η απόφαση πρέπει να πάρθει από τις Ιρλανδικές Αρχές. Το άρθρο 172 για τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάει γι' αυτό. Έχει λόγο η Ιρλανδία προφανώς για τις υποδομές αυτές. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να σας μεταδώσω σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χάρκιν, ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, θα σύντομη γιατί θέλω όλοι να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Ακούγοντα την προηγούμενη αναφορά, οι πολίτε έρχονται εδώ ότι πιστεύουν ότι υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με τι χωματερέ και θέλουν ε, να ενημερώσουν και να εφαρμοστεί δικαιοσύνη. Εδώ μίλησαν για έλλειψη δικαιοσύνης και δικία. Εγώ διάβασα ε, την απάντηση της Επιτροπής ε, τώρα το ότι υπάρχει υπάρχει ουσιαστικά ε, περιορισμένη χρησιμοποίηση των κονδυλίων στην περιοχή για τη 2000-2006. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις γιατί 10 φορές ε, δαπανήθηκαν κονδύλια σε άλλη περιοχή έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα πραγματικά να δω αυτές τις πληροφορίες που μας είπε η Κομισιόν, γιατί δεν μπορούσα να, βρω, τις βρω τώρα σε ό,τι αφορά το δυτικό διάδρομο σιδηροδρόμων. Βγήκε από αυτό το πρόγραμμα. Πού πήγαν όμως αυτά τα χρήματα, γιατί και αυτό είναι τμήμα των μειωμένων δαπανών. Επίσης, η Κομισιόν αναφερθήκε στο Ταμείο Συνοχής και είπε ότι το Ταμείο Συνοχής, μάλλον η της είπε ότι οι δαπάνες ε, προήρθαν από περιφερειακά ταμεία. Φυσικά το ταμείο συνοχή, τα ταμεία συνοχή είναι εθνικά ε, κονδύλια, όμως η Ιρλανδία μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία συνοχή ε, για το ΕΠ στην λόγω περιοχή ήταν πολύ ε, κατώτερο και έτσι επηρέασε όλο το μέσο όρο και μπόρεσε η Ιρλανδία να έχει πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Έτσι λοιπόν αυτό σας ε, λέει ποια ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης και έτσι λοιπόν εγώ θα ήθελα να δω τη λεπτομερή ανάλυση που έχει η Κομισιόν και τέλος ε, δεν έγινε ανάλυση κόστους ωφέλους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ε, και αν δείτε τα project, ε, ε, κανένα από τα έργα για τα οποία έκανε τη κυβέρνηση ήταν σε αυτή την περιοχή BMW. Όμως εγώ θέλω να δω τις, τα λεπτομερή στοιχεία της Κομισιόν γιατί θα πρέπει να δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια. Πρόεδρος, μάλιστα. Κύριε Άντερσον. Μικρόφωνο παρακαλούμε. οι αναφέροντες αναφέρθηκαν στην αδικία και την έλλειψη διαφάνειας. Ε, είναι αλήθεια ότι αποφάσεις λαμβάνονται στο Δουβλίνο και στο Μπέλφαστ και στην Κομισιόν τους είπαν ότι έγιναν επενδύσεις σε δύο περιφέρειες. Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβαν και ε, τους είπαν ε, ότι στην περιοχή ε, BMWD και στην νοτιοανατολική περιοχή υπήρχαν περιορισμένες κατανομές, όμως αυτό δεν υλοποιήθηκε, αυτά τα κονδύλια δεν δαπανήθηκαν στην περιοχή BMW. Νομίζουμε ότι πρέπει να διερευνηθεί αυτό η West ε, ε, on Track ε, έκαναν έρευνα για αυτό το ζήτημα και σε ό,τι αφορά τα σχόλια της Κομισιόν για κάποια διαβούλευση, ότι έλαβε χώρα κάποια διαβούλευση, όλοι καταλαβαίνουμε πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ διαβούλευσης και δημόσιας διαβούλευσης. Δηλαδή το ότι υπόθηκε ότι υπήρχε μια κάποια διαβούλευση δεν πήθη κανένα. Νομίζω εδώ ότι έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία ε, που σας δίνουν τη δυνατότητα να το διερευνήσετε περαιτέρω αυτό το ζήτημα. Να έχουμε τα στοιχεία που έρχονται την Κομισιόν. Δύο λεπτά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή των Αναφερόντων που θεώρησε ότι είναι παραδεκτή αυτή η αναφορά. Πρέπει να δείτε το χαρτί της Ιρλανδίας. Είμαστε η πλέον απομακρυσμένη και απομονωμένη περιοχή. Επόμενο βήμα, το επόμενη στάση είναι η Νέα Υόρκη. Και όπως είπε η κυρία Χάρκη, είναι τα χρήματα που δόθηκαν για τα διαφορετικά ταμεία, από τα ταμεία συνοχής και όλες τις διάφορες κατηγορίες δόθηκαν όλα στην Ιρλανδία ε, λόγω του ότι το ΑΕΠ μα ήταν ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Όμως πήγαν τα χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών στο Δουβλίνο, τα ξόδεψαν αυτοί όπως ήθελαν και η δική μα περιοχή δεν θεωρήθηκε ως το ένα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σα και μετά όσο είπε η Κομισιόν, ε, γιατί η Κομισιόν μα είπε ότι δεν υπήρχε δημοσία δεβούλευση το 2006 όμως υπήρξε, μετά το 2006, δημοσιοδηβλήψη. Εγώ θα ήθελα να ξέρω πώς ήταν αυτή η δημοσιοδηβλήψη και κάτι που ανέφερε η κυρία Χάρκιν, η Κομισιόν, είπε ότι αν χρειαστούμε θα μας δώσουν λεπτομερή κατανομή. Ναι, τη χρειαζόμαστε. Και κάτι ακόμη. Ε, έγινε σαμποτάζ σε αυτό το Western Track από τους ε, ίδιους τους Ιρλανδούς. Εγώ είμαι το μόνο μέλος της Επιτροπής Μεταφορών της Ιρλανδίας και μπορώ να σας πω ότι η έμφαση δίνεται στους σιδηροδρόμους και παρόλο που είχε εγκριθεί να υπάρχει ένας πλήρης διάδρομος, τελικά το σαμπόταρε η Ιρλανδική κυβέρνηση και η διαφάνεια, βέβαια τίθεται θέμα διαφάνειας, γι' αυτό ήρθαν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι πολύ καλά παρουσιάστηκε η όλη υπόθεση και θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου Πατ Κομπ Γκάλαχερ. Είχαμε μια διαβούλευση στην Ιρλανδία που μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνθηκαν ε, στο Ευρωπαϊκό, ε, στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν ο κ. και σήμερα ε, έχει άλλες υποχρεώσεις και έτσι λοιπόν θα ήθελα να δικαιολογήσω την απουσία του εδώ. Μάλιστα, πιθανότατα θα πάμε το Σεπτέμβριο στην Ιρλανδία και ίσως θα επισκεφτούμε και αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Μάλιστα, θα το σχεδιάσουμε. Σας ευχαριστώ. Ως Επιτροπή θα γράψουμε μια επιστολή, θα συντάξουμε μια επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών. Στον Υπουργό Μεταφορών, με συγχωρείτε. Κύριε Φρέντ. The last issue για το τελευταίο σημείο, την τελευταία αναφορά. Κύριε Πρόεδρε, από τα μελικοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σήμερα εκπροσωπώ τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών όσο και από τον αναφέροντα την Ευρωπαϊκή Ένωση δυσλεξικών. Είμαι ο Christopher Friend και είμαι 100% τυφλός. Στις μέρες μας, σύγχρονο λογισμικό και μαγνητοφορημένα βιβλία μου επιτρέπουν να διαβάζω οποιοδήποτε βιβλίο. Όποιο βιβλίο μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Διότι δυστυχώς 95% όλων των βιβλίων που εσείς μπορείτε να διαβάσετε δεν υπάρχουν σε μορφή διαθέσιμη για τυφλούς όπως εγώ ή για άτομα με δυσλεξίες όπως ο κ. Κάμερο ο οποίος κάθεται δίπλα μου. Ακούσατε από προηγούμενε παρεμβάσει μα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών που εκπροσωπεί 285 εκατομμύρια ανθρώπων με προβλήματα ώρες εναν τον κόσμο έχει ξεκινήσει μια σχετική εκστρατεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματική Ιδιοκτησίας. Εάν τροποποιηθεί ελαφρώς η σχετική νομοθεσία θα επιτρέψει στους ανθρώπους τους δυσλεξικούς αλλά και με προβλήματα όρασης να αγοράσουν και να στείλουν βιβλία πέρα από σύνορα. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει η σχετική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέλη της Φοιτοποίησης θα θυμούνται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσαν σκληρή μάχη να μπλοκάρουν τη συνθήκη για τους τυφλούς. Πέρσι όμως χάρη στη δική σας βοήθεια η Κομισιόν και το Συμβούλιο άλλαξαν θέση και πλέον έχουν εντολή να διαπραγματευτούν μια συνθήκη σχετικώ. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη λύπη, πρέπει να αναφέρω στην Επιτροπή σας ότι οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισαν. Ακόμη και την τελευταία εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα στην Γενέβη. Σύμφωνα με τα πρακτικά, συνέχισαν να επαναλαμβάνω, να επιμένουν να περιληφθεί στο κείμενο της συνθήκης η επέτηση των ιδιοκτών των δικαιωμάτων μια θέση που εξυπηρετεί ακριβώ το λόμπι των εκδοτών. Γι' αυτό Είχε ως αποτέλεσμα ένα κείμενο 9 σελίδων, το κείμενο των 9 σελίδων που είχαμε υποβάλει το 2009, ως Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών, να γίνει ένα τέρας 22 σελίδων, με αναφορές σε ένα σωρό άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που δεν προσφέρει εναλλακτικές ε, λύσεις. Και όλα αυτά για να δικαιολογήσουν την πρότασή του να συμπεριληφθούν επιπλέον διατάξει στην ε, συνθήκη. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν διαπραγματευτέ επικαλούνται την ανάγκη συγκερασμού των δικαιωμάτων των εκδοτών και των δικαιωμάτων των δυσλεξικών και, προβλημάτων, και ανθρώπων με προβλήματα όραση και, και άλλων κατηγοριών ανθρώπων. Τι είδου συγκερασμό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σχέση έχει ο κόσμος των πνευματικών δικαιωμάτων με τα δικαιώματα των τυφλών. Όλες οι σχετικές συνθήκες ούτως ή άλλως ήδη προστατεύουν τους εκδότες. Αυτό το οποίο τώρα πια χρειαζόμαστε με την νέα αυτή συνθήκη είναι μια μη όντως συγκερασμένη, μια μη ισόρροπη προσέγγιση ώστε να προστατευτούν επιτέλους και οι τυφλοί. Όταν καταργήθηκε κάποια στιγμή επιτέλου η δουλεία, δεν ήταν ποτέ διανοητό να υποστηρίξει κανεί ότι πρέπει να εξορροπήσουμε, να συγκεράσουμε τα δικαιώματα των σκλάβων με αυτά των, με την απόλυση οδήματο ενδεχομένω των πρώην δουλεμπόρων. Επιμένουμε ότι αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει. Πέρα από 22 μήνε, τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 12 άλλε χώρε ανά τον κόσμο κατάστρωσαν ένα κείμενο συνθήκη, ένα σχέδιο συνθήκη. Και υπήρχε μόνο ένα κείμενο σε αγγίλε, επρινδέλον είχαν συμφωνήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε και μερικά ανά τον κόσμο κατάστρωσαν ένα κείμενο συνθηκη ένα σχέδιο συνθηκη και υπήρχε μόνο ένα τμήμα σε αγγίλες από τον οποίο δεν είχαν συμφωνήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε και μερικά άλλα κράτη ανά τον κόσμο στράφηκαν κατά της πλειονότητας στον Βάιπο για να καταδικάσουν ακριβώς την συνδίκη του Βάιπο. Επικαλούμενοι διάφορα πράγματα. Αυτή η αδικία λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την πολιτική αρμοδιότητα να σταματήσουν αυτή την αδικία. Εάν δεν τον πράξουν, η Ευρώπη θα είναι ο κακός της ιστορίας. Έτσι θα την αντιμετωπίσουν οι τυφλοί και οι άνθρωποι με προβλήματα όρεσαν τον κόσμο στους διαδρόμους του Άιπος στη Γενέβη πολλοί μας περιγελούν. Η συνθήκη αυτή εξελίσσεται σε μια συνθήκη που προστατεύει τους εκδοτές εις βάρος των τυφλών. Λοιπόν, πρέπει όλα αυτά να πάρουν τέλος αμέσως. Πρέπει να θεσπίσουμε μια αποτελεσματική απλή συνθήκη έτσι όπως πρότειναν οι κοινότητε των δυσλεξικών και των τυφλών ή και ανθρώπων με προβλήματα όραση. Κύριε Πρόεδρε, να υπενθυμίσω στα μέλη τη Επιτροπή σα ότι μένουν λιγότερο από 8 εβδομάδες πριν ξεκινήσει η διπλωματική διάσκεψη για να συζητήσει τη συνθήκη αυτή στο Μαρακέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπερμηνθεί των δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών Λαών και των δικαιωμάτων των τυφλών. Έχετε ρόλο να διαδραματίσετε εν ώψη της έγκρισης στο Μαρακές και πριν την έγκριση βεβαίω στην Ευρώπη. Απευθύνω έκκληση σε όλα τα μέλη τη επιτροπή, μια έκκληση προς όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκήσουν την επιρροή τους στου διαπραγματευτέ, ώστε να κάνουν ό,τι μπορούν για μια απλή συνθήκη υπέρ των τυφλών. Θα είναι μια συνθήκη η οποία θα είναι υπέρ των δυσλεξικών, υπέρ των τυφλών και υπέρ των ατόμων με προβλήματα όρεση τον κόσμο. Ευχαριστώ. Many Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρτίν Πράτ από την Επιτροπή. Oh, Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα στους βουλευτές όπως γνωρίζετε και όπως μας υπενθύμισε ο κύριος Φρέντ η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών και η Ένωση Δυσλεξικών προσπαθεί αυτή την συνθήκη με αποφασιστικότητα. Το αίτημα είναι δίκαιο και αυτό είναι και ο λόγο τον οποίο πολλέ χώρε αυτή τη στιγμή ακριβώ συζητούν αυτή τη συνθήκη στον ＷIPO έχουν μάλιστα δεσμευτεί να δυσφαλίσουν ότι οι εθνικοί νόμοι θα περιλαμβάνουν εξαιρέσεις υπέρ των τυφλών. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και διατάξει που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή βιβλίων πέραν των συνόρων υπό ορισμένε προποθέσει. Εμεί είμαστε μεταξύ αυτών των χωρών που υποστηρίζουν το σχετικό δικαίωμα. Σε πολλέ χώρε υπάρχουν ευνοϊκέ διατάξει για του ανθρώπου με προβλήματα όραση. Αυτό όμω πρέπει να λάβει και μια διεθνή διάσταση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διευκολύνουμε την ανταλλαγή βιβλίων σε συγκεκριμένα φορμάτα, επαναλαμβάνω, από και προ χώρε. στι οποίε ε, ιδιαίτερα δεν υπάρχουν αυτά τα βιβλία. Κατά επανάληψη, το θέμα έτσι όπως το έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών είναι σαφέ. Ισότιμη πρόσβαση στα βιβλία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και ταυτόχρονα με όλους τους άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τούτης, δεν είναι μόνη σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν οι ΗΠΑ, μεταξύ άλλων η Βραζιλία, η Ινδία, ο Καναδάς, η Νιγηρία, η Αίγυπτος, η Ιαπωνία, η Αυστραλία. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις αυτού του τύπου, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πολύπλοκες. Δυστυχώ, και παρά του ισχυρισμού ορισμένων ΜΚΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη τη δεν έχει την δύναμη να εγκρίνει την συνθήκη. Κάθε αντιπροσωπεία συμμετέχει με διαφορετικά αιτήματα στι διαπραγματεύσει. Εξού και ανάγκη να διαπραγματευτούμε. Για παράδειγμα, στον τελευταίο γύρο στην Γενέβη, η Αίγυπτο επέμεινε να συμπεριληφθεί στη συνθήκη το δικαίωμα τη μετάφραση. Κάτι το οποίο δεν ζήτησαν καν ποτέ τυφλοί. Η Ινδία ήθελε να συζητήσουμε την ερμηνεία της συμφωνίας TRIPS στο πλαίσιο του WIPO. Οι ΗΠΑ Πολιτείες ήθελαν να παραχωρήσουν όσον αφορά μια συμφωνία που είχαμε επιτύχει το Φεβρουάριο τη σχέση μεταξύ της νέας συνθήκης δηλαδή και τη των διεθνών υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν 8 εβδομάδες πριν την έναρξη της διπλωματικής διάσκεψης είμαστε στον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων είμαστε ακόμη μακριά από τον στόχο μα. Συμφωνώ με την Ένωση Τυφλών ότι το κείμενο είναι υπερβολικά πολύπλοκο, υπάρχουν υπερβολικά πολλέ αγγείλε, πολλά τμήματα του κειμένου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και έχουμε διαφορετικέ προτάσει διατύπωση. Πέρα από τι δικέ μα θέσει υπάρχουν, να ξέρετε, και θέσει και ανάγκε και άλλων χωρών. Αν θέλουμε να πετύχουμε στο Μαρακές, και όταν λέω να πετύχουμε εννοώ να έχουμε στα χέρια μας μια αποτελεσματική συνθήκη η οποία θα ικανοποιεί την ανάγκη πρόσβαση στα βιβλία των τυφλών. Αν θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε πρέπει να προσπαθήσουμε γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δεν θέλουμε μια συνθήκη η οποία δεν θα είναι αποτελεσματική ή μια συνθήκη η οποία δεν θα επικυρωθεί στη συνέχεια. Σε πω μεταξύ της σημερινής ημέρας και του Μαρακές θα προσπαθήσουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας ακόμη και αν δεν είναι προγραμματισμένη σαφώς επίσημη γύρι διαπραγματεύσεων. Και το λεφτό για γιατί στο δεν θα είναι δυνατόν να τα λύσουμε τα πάντα. Τις θέσεις αυτές σημερίζονται οι περισσότεροι γύρω από το τραπέζι που πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο να συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση συμπεριλαμβάνοντας και όλους τους εμπλεκομένους. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, διότι όπως σε κάθε διαπραγμάτευση δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε εάν δεν ικανοποιούμε λίγο πολύ τους πάντες. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Όσο πιο απλό είναι ένα κείμενο, και το ανέφερε αυτό κύριος Friends, τόσο, τόσο πιο εύκολα θα συμφωνήσουμε και θα επικυρώσουμε την συμφωνία μας. Πρέπει λοιπόν στην προσπάθεια να συμπεριλάβω τις πάντες. Η πρόεδρος λέει να τελειώνει η ομιλήτρια. Έχουμε μόνο 15 λεπτά ακόμη που μας έδωσαν διερμηνείς. Λοιπόν, να πω το εξή, λέει ομιλήτρια, μεταξύ αυτής της συνεδρίασης και του Μαρακές θα προσπαθήσουμε να περάσουμε το πολιτικό μήνυμα σε διάφορα επίπεδα, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα πέρα από τεχνικό. Έτσι, στο Μαρικέστο είμαστε έτοιμοι να ξυπνήσουμε τον διαθέσιμο χρόνο. Κύριε Κάσμα, ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και πρέπει να συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση. Συμφωνώ απόλυτα με μας υποθήκαν από τον αναφέροντα. Θα ζητούσα από του διαπραγματευτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συνεχίσουν να προσπαθούν επί αυτού του θέματο και τον το Μισελ του πω ότι τώρα θα σταματήσαμε να ζητάμε διατύπωση για τα άρθρα D e που αφορά την ε, διεθνή την πρόσβαση σε βιβλία και απαιτεί προϋπόθεση ένα βιβλίο να έχει τεθεί σε εμπορία αλλά δεν θα πρέπει πλέον να ζητούνται αυτές οι προϋποθέσεις γιατί αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα και σας προτρύνω Πρόεδρε να ζητήσουμε μια επίγουσα συνεδρίαση με τον κύριο Μπαρνιέ για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ναι, εξαιρετική ιδέα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Λιχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όσα είπατε και να προσθέσω κάτι ακόμη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το να στέλνουμε τα διαθέσιμα βιβλία σε ιδιώτες, γιατί αν περιορίσουμε τα πάντα για τις οργανώσεις των τυφλών, τότε οποιοδήποτε άνθρωπος που ζει στην εξοχή και είναι απομακρυσμένος, το χάρη, δεν θα έχει καμία πρόσβαση στα βιβλία. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο διατάξεις είναι αυτές που πρέπει να διευρυνθούν και να υπερασπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αποτελούν ε, κάτι πολύ σημαντικό γιατί δυσκολεύουν τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν θα ζητήσω να φροντίσετε να ζητήσετε αυτές τις τροπολογίες και κάτι ακόμα. Θα ήθελα εγώ να ε, δω και την εντολή με εμπιστευτικό τρόπο γιατί ε, ήμουν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αλλά μου το αρνήθηκαν αυτό για τη διαφάνεια, για να σχολιάσω το θέμα της διαφάνειας. Καλό. Oh. Ο κίνδυνος ε, εδώ είναι να μην αλλάξει τίποτα. γιατί η προσέγγιση της Κομισιόν ε, και του Μισελ Μπαρνιέ που καταρχήν ήταν εχθρική ενώ τώρα έκαναν το πάρα πολύ σημαντικό βήμα να επιμένουν για αυτή τη συνθήκη ο κίνδυνος ε, είναι οι δυσκολίες που μας ε, ανέφερε η κυρία Πράτ και εγώ την πιστεύω, πιστεύω το είπε να μην επιτρέψουν να έχουμε ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ένα πρακτικό πλεονέκτημα, ε, την, ε, το πολιτικό όφελος του να έχουμε τη συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρεωθεί μια ουσιαστική αποτυχία Αλλιώς ε, πρέπει να επιμείνουμε για τα άρθρα D και E. Θα πρέπει να καταργηθούν ε, αυτά τα αυτές οι γραφειοκρατικές διατάξεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να είμαστε ε, πολύ πιο κάθετοι, να αντισταθούμε στις δυσκολίες που μας θέτουν οι άλλοι διαπραγματευτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα γιατί δεν θέλουμε μόνο να διευκολύνουμε την εμπορική διαθεσιμότητα γιατί η κυκλοφορία των βιβλίων, μπορεί να, η διακίνηση των βιβλίων μπορεί να γίνει και μέσω άλλων μορφών, μέσω βιβλιοθηκών παραδείγματο χάρη. Δεν μπορεί τώρα εδώ να απαιτούμε προπόθεση να υπάρχει μια οργάνωση που να διασφαλίζει τη δυνατότητα του τυφλού να έχει πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στην Επιτροπή Νομικών Θυμάτων όπου συζητήσαμε το copyright, αυτό το πρόβλημα του copyright και της μη εύκολης ε, πρόσβασης είναι το αποτέλεσμα ενός εγωισμού κάποιου που θέλουν να ε, υπερασπιστούν κάποια πλεονεκτήματα του copyright. Όμως εδώ αυτά που συζητάμε έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο κάθετοι στις διαπραγματεύσεις. Ε, Mrs. I simply would like to add πολύ σύντομα να προσθέσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι ώστε να εξακολουθούμε να θυμόμαστε περί τίνος πρόκειται. Πάει κανείς σε μια βιβλιοθήκη όλοι μας, εκτός από τους ανθρώπους με προβλήματα όρεση, μπορεί να διαλέξουν από τα βιβλία που υπάρχουν στο ράφι, ενώ οι άνθρωποι με προβλήματα όρεση μπορούν να διαλέξουν μεταξύ πέντε βιβλίων. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό εννοούμε ως ελευθερία. Δηλαδή εγώ συμφωνώ με όλα όσα είπατε και τα υποστηρίζω. Απλά να μας υπενθυμίσω πώς ε, έχουν τα πραγματικά γεγονότα, γιατί πράγμα συζητάμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν ε, τους μεταφραστές ότι μας έδωσαν λίγο τόση ώρα παραπάνω. Να πω ότι πέρα από την πρόταση του κύριου Κάσμαν να, για μια συνάντηση με τον κύριο Μπαρνιέ, μια ε, προφορική ερώτηση στη διάρκεια της ολομέλειας που να αφορά το συγκεκριμένο θέμα από τη μεριά της επιτροπής νομίζω ότι επίσης θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση που επισημάνατε. να είστε καλά ευχαριστώ και τους ε, ε, αναφέροντες που ήταν εδώ και μας έδωσαν δυνατότητα να σκεφτούμε. Κοιτάξτε, κάποιες ομάδες ήθελαν να, θέσουν προφορική ερώτηση. Τουλάχιστον ε, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες είχαν υποστηρίξει αυτήν την ιδέα. Υπάρχει προφορική ερώτηση με απάντηση στο Στρασβούργο. Μάλιστα, ευχαριστώ.